So, good afternoon, everybody. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στην απογευματινή συνεδρίαση τη Επιτροπή ΣΥΜΚΟ, Συντροφή Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών. Με μεγάλη χαρά ε, καλωσορίζω εδώ τον Ρίτσαρντ Μπρούτον, που είναι Υπουργό Εργασία, Επιχειρήσεων και Καινοτομία. Φοβερό τίτλο. Είναι τόσο σημαντικά αυτά τα χαρτοφυλάκια, είναι φοβερό να είσαι υπεύθυνο. Χρειαζόμαστε περισσότερα από όλα. Περισσότερε θέσει απασχόληση, επιχειρήσει και καινοτομία. Ε, ο πρόεδρο ε, του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα επίση θα μα ενημερώσει για αυτά. Θα ήθελα να κάνω δύο-τρει αναγγελίε ε, πριν ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να σα πω ότι περνάμε στο διαδίκτυο. Ελπίζω να μας παρακολουθούν πολύ παντού και πολύ στην Ιρλανδία γιατί είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για τη συνεργασία που θα έχουμε με την Ιρλανδική Προεδρία το επόμενο εξάμεινο. Ε, μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο γιατί είσαστε υπεύθυνοι και θα, για διάφορα θέματα που εμείς θέλουμε να προωθηθούν. Ένα μέλος Ιρλανδός της Επιτροπής μας ε, ενδιαφέρεται πολύ για αυτά τα θέματα. Επίση, πίσω στην αίθουσα ε, υπάρχει μια ομάδα από φοιτητέ από το Πανεπιστήμιο Άστον ο Νατάλιαν Κόψε και η Καρολάιν Ρο είναι επικεφαλής αυτής της ομάδας ε, και είναι τμήματα ενός ε, σημαντικού ερευνητικού Ινστιτούτου. Αυτοί έχουν φέρει αυτούς τους φοιτητές. Ε, ήρθαν εδώ για να παρακολουθήσουν στην πράξη τι κάνουμε εμείς. Σας καλωσορίζω στην συνάντησή μας, λοιπόν. Ο Ρίτσαρτ Μπρούτον είναι επικεφαλής τώρα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, είναι ο Προεδρεύων. Είναι άτομο με μεγάλη κατανόηση για την δική μας τη δουλειά και πιστεύω ότι θα προχωρήσει αυτά τα θέματα. Του δίνω το λόγο για να μας πει δύο λόγια για τις προτεραιότητες της Προεδρίας του και να μοιραστεί τις σκέψεις του μαζί μου, μαζί μας. Και βεβαίως έχω και έναν ανοιχτό κατάλογο μιλητών για οποιονδήποτε θέλει να υποβάλει ερωτήματα. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, Ρίτσαρντ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Μάλκομ. Νομίζω ότι η δουλειά σας έχει κάνει εξαίρετο έργο και για μένα είναι πολύ καλή ευκαιρία που μπορώ να έρθω εδώ και να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Γνωρίζω ότι από την προηγούμενη φορά πριν από 15 χρόνια που είχα έρθει, από τότε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικά τα θεσμικά όργανα έχουν γίνει πολύ πιο δημοκρατικά. Εκτιμώ όλους ιδιαίτερα στο ρόλο που έχετε παίξει εσείς και τους βλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία μαζί σας στα διάφορα θέματα για τα οποία θα συνεργαστούμε. Η ενή αγορά, αναμφίβολα, αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για μας είναι ένας ε, τομέας στον οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε και να έχουμε πιο ισχυρές οικονομικές σχέσεις μεταξύ μας. Ξέρω ότι η δικιά σας προεδρία ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή προκειμένου η αλλαγή αυτή να γίνει. Τώρα, το γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης όπου βρισκόμαστε, είναι πολύ βασικό να ξανασκεφτούμε τη λογική δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δείχνει τι ε, δεσμοί υπάρχουν μεταξύ των χωρών μας και ότι υπάρχουν κοινοί κίνδυνοι τους οποίους ε, συμμεριζόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουν μαζί τις δυσκολίες μέσα από μια συνένεση και μέσα από το σεβασμό της διαφορετικότητας. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πάρα πολλέ φορέ και έχω διαπιστώσει ότι εσεί προχωράτε προ αυτή την κατεύθυνση, Πρόεδρε. Τώρα, η οικονομική ανάκαμψη, η ε, βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, απαιτούν ε, την κατάργηση των εμποδίων. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να λειτουργήσει ανεμπόδιστα και με δυναμισμό η ενιαία αγορά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2012 με τα συμπέρασμά του ζητάει από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουν στην ε, πράξη, την πρώτη πράξη της ενιαίας αγοράς και να προχωρήσει σε θέματα όπω είναι τα επαγγελματικά προσόντα, οι δημόσιες συμβάσεις και η απόσπαση των εργαζομένων. Η εσωτερική αγορά λοιπόν έχει πολλά ωφέλη για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να δώσει όθηση και στην οικονομία της. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταργηθούν όλα τα ενδοευρωπαϊκά εμπόδια στο εμπόριο που υπάρχουν Κάτι το οποίο το κάναμε βέβαια τα τελευταία χρόνια και αυτό φάνηκε από μια αύξηση 14% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλεται ακριβώς στην ελευθέρωση αυτή του εμπορίου. Σήμερα που οι χώρες μας ε, υποφέρουν όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, είναι σαφές ότι ο δυναμισμός πίσω από αυτή την ευάθμιση της νέας αγοράς στην Ευρώπη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να διευκολύνω συμφωνίε μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με την πράξη για την ενία αγορά 1. Η νομοθεσία τώρα για την ενιαία αγορά επίσης πρέπει να αποκρίνεται στα κριτήρια της τεχνολογικής πρόοδου που έχει επιτεθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Πρέπει να μειωθεί το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για παράδειγμα και να υπάρξει καλύτερη προστασία και διευκόλυνση μετακίνηση διεθνώ των εργαζομένων. Η Ιρλανδική Προεδρία πρόκειται να ελέγξει και να παρακολουθήσει την πρόοδο που έχουμε με την, για όλα τα θέματα της ενίας αγοράς και ιδιαίτερα θα αναφέρεται στην Κορεπέρ και στο Συμβούλιο. Με τέτοιου είδους διαχείριση των ε, θεμάτων η Προεδρία πιστεύει ότι θα μπορέσει χωρίς κλειδονισμούς αλλά και αποτελεσματικά να ανταποκριθεί ε, στα αναδιόμενα και στα νέα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Ιδιαίτερα πρόκειται να ασχοληθούμε και να συνεργαστούμε μαζί σας όσον αφορά το πακέτο για τις δημόσιες συμβάσεις, το, σε ελέγχους λογαριασμών, τα μέτρα λογιστικού ελέγχου και άλλες προτάσεις για την εμβαία αναγνώριση των προσόντων και την απόσπαση των εργαζομένων. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ για ό,τι έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και θα προσπαθήσουμε στην πράξη, στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, να προωθήσουμε περισσότερα θέματα. Μόνο αγκαλιάζοντα την ψηφιακή επανάσταση μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ελπίσει ότι θα αντιμετωπίσει σφαιρικά τον 21ο αιώνα. Η ανάπτυξη τη ψηφιακή οικονομία επίση θα προωθήσει το διασυνοριακό εμπόριο και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, ε, δίνοντα ε, μακροπρόθεσμα ωφέλη και στι επιχειρήσει και στου καταναλωτέ. Θα συνεχίσουμε επίση με προθυμένα μέτρα όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά προκειμένου να υπάρξει εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές συναλλαγές σε τομείς όπως είναι η ηλεκτρονική υπογραφή, όπως επίσης θέλουμε να προχωρήσουμε και σε θέματα ε, του πακέτου πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνουν την οδηγία copyright και την συλλογική ε, διαχείριση ε, δικαιωμάτων. Κάτι το οποίο έχει να κάνει με την αδειοδότηση συγχρόνως σε διαφορετικές χώρες για την διανομή online μουσικών έργων. Είναι πολύ βασικά όλα αυτά για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Πρέπει να λυθούν τα διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το copyright και τις αδειοδοτήσεις. Εκ παραλλήλου, στο νομοθετικό έργο προτείνουμε οι Υπουργοί να συζητήσουν στο Συμβούλιο τον Μάιο για το θέμα των αδειών στην Ευρώπη, που είναι ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επίσης και για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις, προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια ψηφιακή ενιαγορά. αγορά. Θα συνεχίσουμε στο Συμβούλιο να επιταχύνουμε τα σημαντικά θέματα της πράξης της ενιαίας αγοράς, με προτάσεις που περιλαμβάνουν την αναθεώρηση του κοινοτικού σήματος, όπως επίσης και την οδηγία για την προσέγγιση των ε, εθνικών νομοθεσιών για το εμπορικό σήμα. Όπω επίση να κάνουμε και προτάσει για τροποποίηση τη οδηγία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. Επίση, θέλουμε και την επικύρωση τη συμφωνία για το ενιαίο δικαστήριο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία και για την ενιαία ε, προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία και να διακανονίσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την μετάφραση. Ερχόμαστε τώρα στα θέματα δημοσίων συμβάσεων και τη σχετική οδηγία με την αγορά δημοσίων συμβάσεων να είναι υπεύθυνη για το 19% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, η μεταρρύθμιση η σχετική προσφέρει μια πολύ σημαντική ευκαιρία για ανάπτυξη και καινοτομία παντού στην Ευρώπη. Πολύ πρόοδο έχει επιτευχθεί υπό την ε, Προεδρία τη Δανία και την Κυριακή επίση Προεδρία σε σχέση με τι προτάσει για τι δημόσιε συμβάσει και η συμφωνία ε, επιτεύχθη το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Αυτή η συμφωνία ε, που επετεύθη. Επετεύθη μετά από πολλή δουλειά που έγινε σε ομάδε εργασία του Συμβουλίου. Και γνωρίζω ότι και η Επιτροπή σα και οι συγκητέ και οι σκιώδε και αυτοί έκαναν τεράστιε προσπάθειε για να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία όσον αφορά τι δημόσιε συμβάσει ολόκληρη την Ευρώπη. Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο τώρα εξετάζουν τροπολογίες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να δεσμευτούμε ενεργά και να πετύχουμε μια τελική συμφωνία για όλες τις προτάσεις. Για να διευκολυνθεί τώρα αυτή η διαδικασία διαπραγμάτευσης έχουμε ήδη ξεκινήσει άτυπες επαφές μαζί σας και με τους συζητητέ, τον κύριο Ταραμπέλα και τον κύριο Γιουβέν. Η θετική φύση της σχέσης αυτής με κάνει να έχω εμπιστοσύνη για το ότι θα δουλέψουμε σε πνεύμα συνεργασίας για να πετύχουμε τον στόχο μας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ιρλανδίας. Ο εξεχρονισμός και αναγνώριση τώρα των επαγγελματικών προσόντων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχυθεί η κινητικότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για μας μια προτεραιότητα και θα προσπαθήσουμε να βασιστούμε στη δουλειά που έχει κάνει η Κυπριακή Προεδρία αλλά και της Δανίας προηγουμένως. Όλα αυτά βέβαια είναι αρμοδιότητα του συναδέρφου μου Ρούρι Κουίν που μου ζήτησε να σας μεταφέρω ότι δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί σας σήμερα το απόγευμα. Ξέρω όμως ότι έχετε δουλέψει για αυτό το θέμα πολύ και ότι δίνεται μεγάλη σημασία στο να προχωρήσει. Η Προεδρία μας επίσης θέλει να επιτευχθεί συμφωνία για πιο περίπλοκες υποθέσεις. Θα πρέπει να έχουμε κάποιο συμβιβασμό βέβαια μεταξύ των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου για να λυθούν διάφορα ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα. Είμαστε πεπισμένοι όμω ότι η δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα η Επιτροπή σα και ομάδε εργασία του Συμβουλίου θα έχουν σαν αποτέλεσμα να τα καταφέρουμε. Συνεχίζουμε επίση και προσπαθούμε να πετύχουμε μια γενική προσέγγιση για θέματα όπω είναι η έλεγχη λογαριασμών και η λογιστική για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις επίσης και για την απόσπαση των εργαζομένων, τη σχετική δηλαδή οδηγία. Η Ιρλανδία στηρίζει παρετέρω προσπάθειες για να βελτιωθούν οι λειτουργίε και ό,τι έχει να κάνει με την ενιαία αγορά που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί και κινητήρια δύναμη για την ανταγωνιστικότητά τη, την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την κινητικότητα στην Ευρώπη. Ξέρω επίσης ότι προσπαθούμε να πετύχουμε και συμφωνία σε μέτρα τα οποία μάλλον όχι μόνο σε, στην υιοθέτηση μέτρων, αλλά και στην εφαρμογή των μέτρων, να δούμε πώς δηλαδή λειτουργούν αυτά στην πράξη. Και πιστεύω ότι η έκθεση του κυρίου ΣΒΑΠ από ε, αυτού είναι μια έκθεση που συζητήσατε σήμερα και βοηθάει πολύ. Πρέπει βέβαια να μειώσουμε και την περιττή και άχρηστη και βλαβερή ε, γραφειοκρατία πολλέ φορές. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε σε μια νέα προσέγγιση για τα καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με νέα μεθοδολογία προκειμένου να έχουμε ευφυεί ρυθμίσει και νομοθεσία. Έχει ήδη επιτευχθεί πρόοδο σε σχέση με αυτά σε συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα το μέλλον. Για τον ε, τελωνιακό κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίση η Προεδρία μα θέλει να πετύχει συμφωνία με το Κοινοβούλιο και να διασφαλίσει την έγκριση της σχετική πρότασης. Τώρα έρχομαι στα θέματα καταναλωτών, ιδιαίτερα την προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση των δικαιωμάτων του. Η πρόταση που έχουμε όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για την ε, ασφάλεια των προϊόντων τώρα και τα μέτρα αποπτία της αγοράς είναι πολύ σημαντικέ πρωτοβουλίες που θέλουμε να προχωρήσουμε κατά τη διάρκεια της Ελλαδικής Προεδρίας. Πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουν συζητήσεις επί των υποθέσεων αυτών για να ασφαλίσουμε ότι θα ολοκληρωθούν σε συνεργασία βέβαια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την άνοιξη του 2014. Τέτοιες προτάσεις έχουν να κάνουν με την καρδιά των πραγμάτων που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές μας, έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των καταναλωτών ιδιαίτερα μάλιστα φέτος που είναι η χρονιά του πολίτη και στα πλαίσια επίσης της ε, τρέχουσας οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουμε όλοι. Υπό Ιρλανδικής Προεδρίας επίσης θα συνεργαστούμε στενά με το Κοινοβούλιο για να ολοκληρώσουμε το έργο μας για το πρόγραμμα των καταναλωτών, που αποτελεί βάση για την εφαρμογή της ατζέντα των καταναλωτών, που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική όπως και εσείς. Τέτοιοι στενοί δεσμοί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια ε, βοηθούν επειδή το κλίμα μέσα στο οποίο συνεργαζόμαστε είναι πάρα πολύ θετικό και το ξέρουμε αυτό και από την μελέτη που κάναμε των νέα ε, τεχνικών οδηγιών με την απόφαση 768 του 2008 στο πακέτο για την τεχνική εναρμόνιση. Επίσης ε, θέλω να σας πω ότι εκτιμώ όλου ιδιαίτερω τι καρποφόρες συζητήσεις που είχαμε με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπό Κυπριακή Προεδρία για θέματα που έχουν να κάνουν με την οδηγία εναλλακτικών τρόπων επίλυση διαφορών και την online επίλυση διαφορών, κάτι το οποίο για το καταναλωτή είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι οι προτεραιότητε αυτέ οι οποίε δείχνουν πόσο μεγάλη σημασία δίνει η Ιρλανδία στο να δημιουργηθούν οι κατάλληλε συνθήκε και το περιβάλλον στην Ευρώπη ώστε να προωθεί η απασχόληση, η ανάπτυξη και να βαθύνουμε ακόμα περισσότερο στην ενιαία αγορά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα, κύριε Πρόεδρε. Good. Okay, well... λοιπόν. Ε, Μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα τα μέλη. Έχουμε πολλούς σημαντικού φακέλους φυσικά εδώ και θα ήθελα να καλέσω την κυρία Πέντρικα στο πολύτιμο και μέλος της Επιτροπής μας. Ας ακούσουμε πρώτα δύο ερωτήσεις και μετά είμαι σίγουρος ότι οι συντονιστές, ο κ. Μάντερσον, ο κ. Σουάμπ θα θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Α ακούσουμε πρώτα την κυρία Πέτρικα και την κυρία Κόλας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Δεν θα ξεκινήσω κάνοντα μια ερώτηση. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία το να καλωσορίζουμε τον Υπουργό στην Επιτροπή μα. Είναι πολύ σημαντική η Επιτροπή μας, έτσι πιστεύουμε όλοι εδώ. Φυσικά είναι πολύ διαφοροποιημένη και επικοινόμορφη η Επιτροπή μας και δεν είναι εύκολο να εστιαστούμε μόνο σε μία πτυχή. Θα ήταν σαν να υποβαθμίζουμε το έργο που κάνουμε σε όλα τα υπόλοιπα θέματα. Είναι τεράστια ευκαιρία για εμάς ε, το ότι μπορούμε να σας δείξουμε ένα κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε εδώ στην Επιτροπή μας και τι εξωτερικές επιπτώσεις έχει. Θα επανέλθω με ερωτήσεις αργότερα, αλλά θα ήθελα ως το μόνο ε, μέλος από την Ιρλανδία να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας και να αφήσω τους όσους ε, έχουν ε, δουλέψει σκληρά ως Ήγητες ε, να ξεκινήσουν τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Uh, Κυρία Κοράτσα Μπέλτ, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον Υπουργό. Αυτές οι προτεραιότητες για τη σταθερότητα και τις θέσεις εργασίας ε, είναι προτεραιότητες και για εμάς. Θα ήθελα να θέσω ειδικότερα σε εσάς το ζήτημα της οδηγίας για τις υπηρεσίες, την ψηφιακή Ευρώπη και τη λιανικό εμπόριο. Εγώ είμαι εισηγήτρια της εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες. Όπω ξέρετε το συζητάμε ήδη εδώ και καιρό. Ε, και έχουμε, υπάρχει κίνδυνος λάθος εστίασης και κόπωσης. Οι προσδοκίες ήταν είναι υπερβολικά υψηλές για τις θέσεις εργασία. Θα χρειαστεί να μειώσουμε τι προσδοκίε, λέμε. Και η γραμμή που θα ήθελα να ακολουθήσω εγώ και ελπίζω να συμφωνήσουμε γι' αυτό είναι η εξή. Η δυνατότητα τη δημιουργία θέσεων εργασία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, χωρί να ξοδεύουμε τα λεφτά των φορολογουμένων, βασίζεται στη σωστή υλοποίηση τη οδηγία για τι υπηρεσίε. Μπορούμε να συνεχίσουμε να την ερμηνεύουμε, αλλά δεν χρειάζεται να την αλλάξουμε. Μπορούμε να την προσαρμόζουμε φυσικά βάσει των προόδων των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των ε, υπηρεσιών. 17 επιστολές προειδοποιητικές έχει στείλει κομισιόν στα κράτη-μέλη και θα ξεκινήσει η διαδικασία κατά 11 κρατών μελών. Δεν χρειάζεται να ε, επινοήσουμε ξανά τον τροχό. Απλά πρέπει να βάλουμε τον τροχό σε κίνηση. Είναι τεράστια ευθύνη. Σκεπτόμενοι ότι τόσο μεγάλο κομμάτι της ψηφιακής οικονομίας βασίζεται στις υπηρεσίες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να θέσετε το ζήτημα της σωστής και πλήρους υλοποίησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες και την αντιμετώπιση των κρίσεων ζωνών, διότι διάφορα κράτη-μέλη την έχουν εφαρμόσει σε διάφορα επίπεδα, σε επίπεδο δήμων, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει υλοποιηθεί, αλλά υπάρχουν κρίσεις ζώνες. Και το να στερούμε θέσεις εργασίας από τους πολίτες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή Πραγματικά ελπίζω να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πολιτική σας αποφασιστικότητα και τη θέση σας για να προχωρήσουμε με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την υλοποίηση, την επιβολή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Επίσης, εγώ ήμουν εισηγήτρια για το τομέα του λιανικού εμπορίου. Η Κομισιόν τώρα ε, σχεδιάζει ένα σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο. Ε, το έχουμε συμπεριλάβει στην πολιτική ατζέντα μακροπρόθεσμα για πρώτη φορά μιλάμε για πάνω από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν ε, προτίθεστε να το θέσετε σε ένα το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας υπό την Προεδρία σας ώστε να υπάρξει αυτή η μακροπρόθεσμη επικύρωση και από τα κράτη-μέλη. Κάτι που προς το παρόν έχουμε επιτύχει σε κάποιο βαθμό χάρη στην εξαιρετική συνεργασία και στην ίδια, την ίδια γραμμή με την Κομισιόν. Αυτό το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπίζεται διαρκώς και πρέπει να ε, υλοποιηθεί η βάση μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Το τρίτο σημείο αφορά την ψηφιακή Ευρώπη, το ανέφερα ήδη. Θεωρείτε υπάρχει ενδεχόμενο ήδη κατά την Προεδρία σας να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και πάλι Ναι, έχουμε, προβλέπουμε κάποια εμπόδια ότι υπάρχει, ε, είναι δύσκολο να επωφελούμαστε από τις ε, ε, διασυνοριακές online υπηρεσίες φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας αφήσω κύριε Υπουργέ να απαντήσετε και μετά θα ακούσουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Καταρχάς σας ευχαριστώ που θέτετε το θέμα της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες. Συμφωνώ με την άποψή σας ότι οι πιο σημαντικές ευκαιρίες είναι η εφαρμογή της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες και την ενιαία αγορά και οι συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου. Χαίρομαι που η Κομισιόν δουλεύει σε αυτό το τομέα. Έχει εντατικοποιήσει τη δουλειά τη με τα κράτη-μέλη. Ε, συναντιόμαστε σε ομάδες, ε, κάνουμε αξιολόγηση ομοτήμων και ε, εξετάζουμε τις προειδοποιητικέ επιστολές αυτές και ενδέχεται να προβούμε και σε άλλες διαδικασίες επί παραβάση. Σίγουρα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή, λέει το Συμβούλιο, στα ορόσημα ανταγωνιστικότητας. Πρέπει να δούμε την πρόοδο εφαρμογής με συστηματικό τρόπο. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο ρόλος του καθενός στη διαδικασία. Συμφωνώ με σας ότι εδώ θα πρέπει να προχωρήσουμε και θα υποστηρίξουμε την Κομισιόν στην δουλειά της. Για το σχέδιο δράσης για το λιανεμπόριο. Άκουσα αυτά που είπατε σε αυτή τη φάση δεν έχουμε προβλέψει τίποτα, αλλά θα το εντάξουμε στις συζητήσεις. Στην οικονομία μας και τη δική μας υπάρχει αντίστοιχη εστίαση στο λιονεμπόριο. Έχει επηρεαστεί πολύ αυτός ο τομέας, υπάρχουν πολύ έντονες τεχνολογικές αλλαγές και θα πρέπει να πάρουμε θέση ούτως ώστε να καταστήσουμε βιώσιμο αυτόν τον τομέα. Υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες στον ψηφιακό τομέα. Θέλουμε να προωθήσουμε τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Ε, στην δεύτερη πράξη για την ενιαία αγορά θα την προωθήσουμε και αυτή. Τις, ε, τα κείμενα για τις προμήθειες με ηλεκτρονικές υποβολές ε, θέλουμε να τα προωθήσουμε. Έχουμε ξεκινήσει στον τομέα του copyright τη δουλειά μας, έχουμε ξεκινήσει τις σχετικές μεταρρυθμίσεις. Είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά και διαιρούν τους εμπλεκόμενους. Ακούστηκαν απόψεις διαφορετικές. Άλλα λένε οι χρήστες, άλλα λένε οι κάτοχοι των δικαιωμάτων. Ούτε οι χρήστες, ούτε οι δημιουργοί περιεχομένου μπορούν να αυξήσουν από μόνοι του τις ευκαιρίες. Θα πρέπει να το κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν θα πρέπει να είμαστε επιτακτικοί ως προς τις αλλαγέ. Αλλά ξεκίνησε η συζήτηση, η Κομισιόν έχει δημοσιεύσει σημαντικά έγγραφα και ελπίζουμε να προωθήσουμε τη συζήτηση και σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Τον Ιούνιο στο Δουβλίνο θα γίνει μια μεγάλη διάσκεψη για την ψηφιακή ατζέντα. Εμείς έχουμε και μία ομάδα για αυτό το θέμα και συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Κουράτσα Μπίλτ για, τον, για το λιανεμπόριο, γιατί εμείς ε, πραγματικά παίζουμε ηγετικό ρόλο εκεί. Ο κύριος Ρόσφορντ θέλει να πάρει το λόγο άλλο συντονιστής, ο κύριος Φαμπ Κέπχαρτ, Μάντερς, κυρία Ρούλε, Πέντεργαρτ, κυρία Ρούλε, επίσης. Λοιπόν, ο κύριος Σβάμπ και η κυρία Γκέμπχαρτ πρώτα, ο κύριος ε, Ρόσφορτ και ο κύριος Μάντες εν συνεχεία. Και στο τέλος η Ιρλανδή κυρία Πέντεγκάρτ Και οποιοδήποτε άλλο ε, ευρωβουλευτή ε, θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Σβάμπ όμως ξεκινάει... Α, παραδίδω τη θέση μου στην κυρία. Κύριε Σβάμπ, σας ευχαριστώ. Σας παίρνω λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας. Αναλαμβάνετε την Προεδρία και βλέπω ότι είσαστε έτοιμος να συζητήσετε θέματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ μαζί μας. Ήμουν ε, εισηγήτρια για την οδηγία για τις υπηρεσίες και επομένως καταλαβαίνετε ότι η εφαρμογή αυτής της οδηγίας με απασχολεί τα μάρλα. Εδώ και τρία χρόνια έχουμε εγγύψει επί της οδηγίας αυτής και ο σκοπός μας είναι να βρεθεί μία λύση στο πρόβλημα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω το εξής. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της οδηγίας. Καταρχάς, πρέπει να σεβόμαστε τα κοινωνικά δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, για να εφαρμοστεί σωστά αυτή η οδηγία. Η οδηγία αυτή Κάθε φορά που συζητάμε την εφαρμογή της, πάντα μπαίνει το οικονομικό θέμα. Τα δικαιώματα των εργαζομένων και η γνώση που έχουν για αυτά τα δικαιώματά τους είναι ένα πρόβλημα που το λησμονούμε συχνά. Θα ήθελα να μας πείτε αν έχετε την πρόθεση να τα θέσετε όλα αυτά, να τα επιθυμήσετε όλα αυτά. Για την εφαρμογή της οδηγίας, ε, Φερρυπίν, έχουμε διαβουλευτεί με τα συνδικάτα, όχι μόνο με τους εργοδότες. Θα πρέπει, αν υπάρχουν πληροφορίες, ή μάλλον να κοινοποιηθούν οι πληροφορίες στους, στις επιχειρήσεις αυτές, για να φτάσουν έως τους εργαζόμενους, γιατί είναι σημαντικές πληροφορίες για τους εργαζόμενους. Ακούστηκε επίσης ότι οι Τσέχοι εργαζόμενοι δουλεύουν στη Γερμανία και τους αντιμετωπίζουν χειρότερα από τους Γερμανούς εργαζόμενους. Έχετε σκεφτεί να θέσετε το ερώτημα αυτό στο Συμβούλιο, γιατί δυστυχώς είναι ένα θέμα το οποίο συχνά το ξεχνάμε όταν γίνεται συζήτηση είτε στο Συμβούλιο είτε αλλού. Ο κύριος Σφάμπ, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Ρίτσαρντ. Σε ευχαριστώ για, την, για τον ενθουσιασμό, για το ζήλο που δείχνεις κατά την ανάληψη των καθηκόντων σου. θέλω εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης να σταθώ και σε αυτά που είπε η συνάδελφος για τις μεγάλες αρχές της ε, εσωτερικής αγοράς. Για αυτές τις αρχές μίλησε και ο Βρετανός Πρωθυπουργό και εκεί φάνηκε η διαφωνία που υπάρχει ανάμεσα στον Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι δομές έχουν θέσει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε σκεφτεί αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν συμβιβασμοί που πρέπει να γίνουν για να λάβουμε υπόψη μας τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Αυτοί οι συμβιβασμοί συχνά αμφισβητούνται από τα κράτη-μέλη. Εγώ ως εισηγητής για την οδηγία για την προστασία των καταναλωτών διαπίστωσα ότι οι συμβιβασμοί που πετύχαμε για κάποιες χώρες ε, αμφισβητούνται σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι απίστευτο, είναι τραγικό. Γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσπαθούμε να επιτύχουμε αυτούς τους συμβιβασμούς. Αλλά τελικά υποσκάπτονται από την ίδια την Ευρώπη. Τους ξεχαρβαλώνουμε με αυτά που κάνουν τα επιμέρους κράτη-μέλη. Θα θέλαμε λοιπόν όλοι μαζί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο Υπουργών να δούμε ποιοι είναι οι μεγάλοι άξονες της πολιτικής για τους καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας θα έχετε πάρα πολλούς φακέλους να, προχωρήσετε, να προωθήσετε. Ας προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Είμαι πεπισμένος ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα κάνουμε και εμείς από πλευράς ΕΛΚ ούτως ώστε να βοηθήσουμε ε, στο να είναι επιτυχής η Προεδρία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό λοιπόν τον κύριο Υπουργό να απαντήσει και μετά θα ακούσουμε τους κύριους Ρόσφαρτ και Μάντρος. Ευχαριστώ πολύ. Υποστηρίζω απόλυτα την απόψή σας ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα πρέπει να έχει ευρεία βάση και θα πρέπει να είναι ισορροπημένη όσον αφορά την εφαρμογή της. Εγώ είμαι μέλος και άλλων ε, σχηματισμό του Συμβουλίου και σκοπεύω να, βρεθώ, να συναντηθώ με τους κοινωνικούς εταίρους και να λάβω και τις απόψεις των συνδικάτων και των εργοδοτών για μια ευρεία απάντηση σε αυτή την ευρωπαϊκή κρίση και για το επόμενο ευρωπαϊκό εξάμενο. Εγώ είμαι λοιπόν ιδιαίτερα υπέρ τη ισορροπημένη εφαρμογή αυτών των κανόνων. Ανοίγουν τι αγορέ, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται με δίκαιο τρόπο. Σαφώς ε, συμφωνώ μαζί σας. Το ενιαίο σημείο επαφής, το single point of contact πρέπει να λειτουργεί δίκαια και όπως έχω καταλαβεί η Κομισιόν έχει αναπτύξει κριτήρια, ορόσημα για αυτά τα ενιαία σημεία επαφής που τώρα έχουν καθιερωθεί και γίνεται έλεγχος της επάρκειας αυτών των κριτήριων. Αυτό θα βοηθήσει, ελπίζουμε, για καλύτερη εφαρμογή και θα ανοίξει περισσότερες ευκαιρίες. Συμφωνώ επίση μαζί σα ότι η διακυβέρνηση τη ενιαία αγορά είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Είχα την ευκαιρία να δω και το δικό σας έγγραφο που έδινε πολύ καλές απόψεις. Πιστεύω το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας υποστηρίζει ιδιαίτερα την άποψη ότι θα χρειαστεί να δουλέψει λίγο πιο σκληρά και να έχει αντίληψη της ανταγωνιστικότητας και της ατζέντα της ενιαίας αγοράς για τα οποία έχει αρμοδιότητα. Αυτή τη στιγμή πιστεύω δίνεται περισσότερη έμφαση στην ε, οικονομική και τραπεζική εξυγίανση ώστε να αντιμετωπιστούν ε, οι μεγάλες προκλήσεις ε, της Ευρώπης. Πολλές όμως από αυτές βασίζονται στην πραγματική οικονομία και στο άνοιγμα των αγορών. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε καλύτερες δομές ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Όπως γνωρίζετε, υπό την Προεδρία μας ε, έχει, δημιουργείται ένα σύστημα αναφορών προς την Κόρεπερ για την πρόοδο των φακέλων της ενιαίας αγοράς. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτό θα βοηθήσει να επικεντρωθούμε στο θέμα περισσότερο. Φυσικά, πρόοδο στους φακέλους προποθέτει συνένεση μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει, θα αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό τώρα τον κύριο Ροσφόρη, συγγητή για το πρόγραμμα καταναλωτών που αναφέρατε και μετά τον κύριο Μάντελ. Κύριε Ροσφόρη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και όλοι μου οι συνάδελφοι κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι εξαιρετική προεδρία για το επόμενο εξάμεινο. Ο δυναμισμός που έχετε ε, δείξει ε, πηγαίνει παράλληλα με την ταχύτητα που, με την οποία ετοιμάζετε το πρόγραμμα σας. Τώρα, μην διαρωτήσω όσον αφορά την οριστικοποίηση του προγράμματος 2014-2020. Έχουμε ήδη συνεργαστεί σε μεγάλο βαθμό με την Κυπριακή Προεδρία αφορούν όλα αυτά. Το επόμενο ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουμε όλοι ότι οι δημοσιονομικές δυσκολίες είναι πολύ σημαντικές. Ε, επίσης ε, θα προβλεφθούν και μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας. Εγώ, συζητητής αυτού του σχεδίου κανονισμού, θα ήθελα να σας πω ότι εάν αποφασιστούν μέτρα δημοσιονομικού περιορισμού, λιτότητας, ελπίζω ότι η Ιρλανδική Προεδρία θα υπερασπιστεί ότι ε, την ε, μη επιρροή του προγράμματος αυτού για τους καταναλωτές, του κονδυλίου για αυτό το πρόγραμμα, για τους καταναλωτές. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της, πολιτικής, της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά πολιτικό θέμα. Σήμερα το πρωί ο κύριος Κάμερον έκανε μια ομιλία στο Λονδίνο που συζήτησε για ένα δημοψήφισμα στο λαό του για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί Θέτω αυτό το ερώτημα εδώ τώρα, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι οφείλουμε στη Μεγάλη Βρετανία πολλά πράγματα όσον αφορά την οικοδόμηση της εσωτερική αγοράς. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε, είναι ένας φάκελος ε, στον οποίο επένδυσε πολλά η Μεγάλη Βρετανία και στον οποίο εργάστηκε σκληρά όπως και ο πρόεδρο τη ε, επιτροπή μα αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο γι' αυτό ο Μάλκομ Χάρμπορ. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή. Ο Βρετανό Πρωθυπουργό φάνηκε να δεσμεύεται για μια έννοια της Ευρώπης αλλά κάρτο, ουσιαστικά λέγοντα ότι η ενιαία αγορά είναι μια χαρά, αλλά ότι τα υπόλοιπα δεν λειτουργούν πολύ καλά. Και ήθελα απλά να σα ρωτήσω, ποια είναι η δική σας θέση, πώς έχετε αναλύσει εσείς το όλο θέμα. Εγώ ως βουλευτής, μέλος αυτής της Επιτροπής, θέλω να πω ότι πιστεύω στην εσωτερική αγορά, πιστεύω ότι αποτελεί μία από τις συνιστώσεις του ευρωπαϊκού οικοδομήματος σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες. Πιστεύω ότι μέσα στην κρίση που βιώνουμε σήμερα χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη. Το ε, κόμμα των φιλελευθέρων στο οποίο ανήκω είναι υπέρ μιας ομοσπονδιακής ε, διαδικασίας προόδου. Αυτό θα βοηθήσει και την ενέα αγορά και ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας άποψη και κατά πόσο συμμερίζετε την ίδια άποψη. Okay, that's an interesting uh, question. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Ε, αυτή η ερώτηση δεν επίπτει ακριβώ στην ατζέντα της Επιτροπής. Φυσικά ε, δεν ξέρω αν ερμηνεύστηκε σωστά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν, έχω προλάβει να την ακούσω. Δεν, θα τη σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Κύριε Μάντερς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και εγώ συντονιστής της ομάδας ALDE ήθελα να σε ευχηθώ καλή τύχη με την προεδρία σας και ελπίζω ότι θα είστε ιδιαίτερα επιτυχείς. Ήθελα και εγώ να μιλήσω λίγο για την ομιλία του Κάμερον σήμερα το πρωί. Αυτός ήθελε ε, ένα, μια διεύθυνση ενιαίας αγοράς αντί για τις διευθύνσεις ε, μεταφορών κτλ. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια διεύθυνση ε, στην Κομισιόν βασικά υπάρχει, αλλά όχι στο Συμβούλιο. Δεν υπάρχει ειδική σύνοδο κορυφή για την ενιαία αγορά, ε, την εσωτερική αγορά. Όλοι μα λένε και το πιστεύουμε ότι η ενιαία αγορά είναι ο πυρήνας τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά παράξενο τρόπο δεν υπάρχει σύνοδο κορυφή για την ενιαία αγορά. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω για όσα είπε ο Κάμερο σήμερα το πρωί. Τώρα, όσον αφορά το Ευρώπη Λακάρτ, δεν σύμφωνα με τα όσα είπε ο συνάδελφο, αλλά καλό θα ήταν να μιλήσουμε για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο. Και αυτό μα φέρνει σε κάτι άλλο. Πέρυσι, τον Οκτώβριο, γιορτάσαμε την Γκράσ. Και μετά από αυτό οργάνωσα μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπή Εμπορίου ε, μία έρευνα με 50.000 ερωτηθέντε, το 68% αυτών των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορούσαν να περιγράψουν, να μας πούν ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς. Κανένας τους δεν είχε ακούσει για το Solvit. Έναν από τον οργανισμό που λειτουργεί άριστα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επιλύει προβλήματα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και του καταναλωτέ. Καμία από αυτέ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν είχε ακούσει ποτέ για το Solvit. Και τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύουμε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για επικοινωνία. Δεν μιλάω για του μισθού των ε, υπευθύνων τύπου που απασχολούμε εδώ, πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία όσον αφορά την ενιαία αγορά. Τι λύσεις θα μπορούσατε να προτείνετε εσείς. Good. Okay. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσω από τον ε, κύριο Υπουργό να απαντήσει στις ερωτήσεις. Έχω και την κυρία Πρέντεργαστ και την κυρία Λεγκρίπ. Αλλά μέλη που θα ήθελαν να σχολιάσουν. Ωραία θα είναι αυτοί οι δύο τελευταίοι ομιλητέ. Α, και ο κ. Κοφεράτη. Δίνω στην κυρία Πρέντερκα. Θα τη δώσω μάλλον τον τελευταίο λόγο, αφού είχε και τον πρώτο. Α ακούσουμε τι απαντήσει προ του συναδέλφου των φιλελευθέρων. Πρώτα απ' όλα, υποστηρίζω και εγώ μαζί σα το πρόγραμμα για του καταναλωτέ. Ξέρω ότι είστε εισηγητή για αυτό. Πιστεύω ότι τα κονδύλια ήταν 170 εκατομμύρια, 197 εκατομμύρια για την περίοδο και σίγουρα είμαστε εμείς ε, διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο για να επιτύχουμε μια συμφωνία. Γνωρίζω ότι εκκρεμούν κάποια ζητήματα, κάποιες διαφορές που θα χρειαστεί να μελετήσουμε, αλλά πιστεύω ότι ο φάκελος αυτός είναι σημαντικός και αναμένω να... τη συνεργασία μας με το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τα ζητήματα Εγώ βρισκόμουν εδώ ω νέο υπουργό στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Τον Λόρτ Κούμπερν ήταν ο, ο κύριο επίτροπο μεταρρύθμιση και αλλαγών. Και αναμφίβολα υπάρχει τεράστια παράδοση Βρετανών βουλευτών που έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της Ευρώπης και στο άνοιγμα των αγορών και στη δημιουργία ευκαιριών εμπορίου και ανάπτυξης. Εγώ φυσικά προερχόμενος από την Ιρλανδία, γειτονική χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, έχω απόλυτη συνείδηση του τρόπου σκέψης του Ηνωμένου Βασιλείου και ε, που οδήγησε και στην ομιλία του κυρίου Κάμερον. Ε, δεν θα σχολιάσω την ομιλία του Πρωθυπουργού μιας άλλης χώρας, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε αυτή την ομιλία πάνω στα οποία θα χρειαστεί να βασιστούμε και ελπίζοντας ότι σε αυτή τη διαδικασία... Η, Βρετανία είναι σημαντικός εμπορικό εταίρο και δικός μας. Ε, ε, μιλάω εδώ ω Ιρλανδός ε, Υπουργός και πιστεύω είναι σημαντικό να προστατεύσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο ως σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως σημαντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά τα σημεία που ανέφερε ο κ. Μάντε, φυσικά η σπουδαιότητα της ενιαίας αγοράς ναι, αποτελεί τον πυρήνα των προσπαθειών μας. Είναι ζωτικό σημείο. Δεν θα πρέπει να διαχωριστεί από άλλα μέτρα. Η Ευρώπη είναι μια ισορροπημένη κοινότητα που προσπαθεί να προχωρήσει σε διάφορα μέτωπα και εγώ αντιλαμβάνομαι τι ευθύνες έχω σε διάφορους τομείς ε, όπως τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί η ισορροπία και θα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ευρώπης που ε, οικοδομούμε. Ε, φυσικά αυτές οι σύνοδοι κορυφής μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση ορισμένων ε, θεματολογίων, αλλά δεν είναι ζωτικό κομμάτι αυτών. Για τα νούμερα που αναφέρετε, το πολύ χαμηλό επίπεδο γνώσεις ε, όσον αφορά τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς, ε, τις χρησιμότητες ενιαίας αγοράς. Αυτό είναι σίγουρα ένα ζήτημα που θα πρέπει να εξετάσει το Συμβουλίο μας. Και είμαι βέβαιος ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντοπίσει τις ελλείψεις ε, όσον αφορά την κοινοποίηση, την ενημέρωση. Τώρα μαζί με τα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο γνωστό στο κοινό το όλο ζήτημα και το να υπάρχει λοιπόν καλύτερη ε, συμμόρφωση και με την οδηγία για τις υπηρεσίες και για την ενιαία αγορά, ε, αυτό θα βοηθήσει να ενημερώνονται καλύτερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις ευκαιρίες που παρέχει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ρίχνουμε φως σε αυτά τα θέματα. Ούτω ή άλλω ζητάμε και από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να δοθεί μεγαλύτερο επίκεντρο στην επικοινωνία. Στην τελευταία έκθεση Gephardt ε, έχουμε συνολικά τρει εκθέσεις για την εφαρμογή της οδηγία για τις ε, υπηρεσίες και έχουμε ε, και μια τέταρτη σκουράτσα build για την πρόθεση. της οδηγία αυτή. Θα ζητήσω από την γραμματεία να σας τις δώσει, ούτως ώστε να πάρετε μια ιδέα. Και ζητήσαμε επίσης ε, να υπάρξουν κέντρα πληροφόρηση στα κράτη-μέλη ε, που θα μοιράζουν φυλά... Α, τα κέντρα μάλλον που υπάρχουν στα κράτη-μέλη να μοιράζουν φυλάδια ε, για την ενιαία αγορά. Δεν λέμε προς πράγματα εμείς στην Επιτροπή μας, τα προωθούμε κιόλα. Η κυρία Γκριπ, ο κύριος Κονφεράτη και τέλος η Ιρλανδή βουλευτής. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Α, θέλει ένα σύντομο σχόλιο, κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Μα σα έδωσα πολύ χρόνο, κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, απευθύνομαι σε εσά επειδή είμαι η συγγήτρια της κοινοβουλευτική αυτής επιτροπής για την αναδιατύπωση του τελωνιακού κώδικα. Χαίρομαι που το αναφέρατε αυτό το θέμα στις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας. Δεν είναι μόνο ερώτηση, είναι περισσότερο μια παρατήρηση, εφόσον μου επιτρέπετε, αυτή που θέλω να κάνω. Σίγουρα γνωρίζετε ότι στα πλαίσια της ιδιαίτερη διαδικασίας αναδιατύπωσης του ενωσιακού τελωνιακού κώδικα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δικιά μας ιδιαίτερη Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει ήδη δουλέψει και ετοιμάσει την εκθεσή της. Γιατί δουλεύουμε ε, με τη λογική προσπαθώντας να τηρήσουμε και τη διαδικασία και τις προθεσμίες. Τη διαδικασία δηλαδή την ειδική για την επαναδιατύπωση. Και έτσι έχουμε ετοιμάσει την έκθεσή μας πριν τα Χριστούγεννα, 17 Δεκεμβρίου ήταν έτοιμη. Αλλά δεν το κρύβουμε από κανέναν βέβαια ότι σε αυτό το στάδιο, από ό,τι φαίνεται, το Συμβούλιο καθυστερεί. Είπατε ότι η ολοκλήρωση της υπόθεσης αυτής αποτελεί προτεραιότητά σας. Όμως, η Ελλαδική Προεδρία, κάνω έκκληση τουλάχιστον, να κάνει ό,τι μπορεί, να πιέσει, να κάνει έκκληση, να συνοδεύσει εντό αγωγικών τα κράτη-μέλη, στο να τα βοηθήσει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και έτσι να μπορέσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να έχουμε τη θέση του Συμβουλίου που περιμένουμε ανυπόμονα θα έλεγα πια. Διότι αν θέλουμε να έχουμε ολοκληρώσει το ζήτημα αυτό μέσα στις προθεσμίες που διαθέτουμε, που είναι πολύ συγκεκριμένες, 24 Ιουνίου φέτος πρέπει να αρχίσει να ισχύει ο νέος κώδικας. Άρα θα πρέπει να κάνουμε όλοι ό,τι περνάει από το χέρι μας, να είμαστε τόσο πιο αποτελεσματικοί, να δουλέψουμε γρήγορα. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο εφόσον έχουμε τη θέση του Συμβουλίου όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και από εκεί και πέρα εσείς με ε, ρεαλιστικό πνεύμα, κύριε Υπουργέ, θα φροντίσετε για την προσέγγιση των απόψεων μεταξύ μας, ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία από την οποία όλοι να έχουν αποφεληθούν, χωρίς να υπερισχύουν τα προνόμια των μεν ή των δε, που να αμβλύνουν το αποτέλεσμα ή να παρακάμπτονται και από την άλλη. Συνεπώς, θέλουμε να χρησιμοποιήσετε την επιρροή σας και να φροντίσετε το Συμβούλιο να έχει κάνει ό,τι πρέπει μέσα στις προθεσμίες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ. Εποφελούμε της ευκαιρίας και της εμπειρίας που έχετε ε, που έχετε και λόγω του χαρτοφυλακίου σας, Υπουργό Εργασίας και Επιχειρήσεων. Για να σας μιλήσω για ένα που μεγάλο πρόβλημα κάτε με για την Ευρώπη του μέλλοντος. Όπως ξέρετε, εμείς ασχολούμαστε με την εσωτερική αγορά. Και ένας, μία από τις προϋποθέσεις για να καταστήσουμε αποτελεσματικό, αποτελεσματικό κάθε τομέα της ενίας αγοράς είναι οι ενιαίοι μηχανισμοί ανταγωνισμού, αναδιανομής του πλούτου, ενιαίοι, μηχανισ... ενιαίοι κανόνες ε, για τις συμπεριφορές ε, των συνομιλητών μας, δηλαδή των Ευρωπαίων πολιτών, ε, όταν λειτουργούν ως καταναλωτές. Οι, κατανα... οι πολίτες, εκτός από πολίτες, ε... και γυναίκες, είναι και εργαζόμενοι. Και ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσουμε συχνά όταν συζητάμε τα θέματα της ε, Επιτροπής μας είναι η έλλειψη ομοιομορφίας στους πραγματικούς και απτούς τρόπους με τον οποίο ε, λειτουργούν οι επιχειρήσεις και από τη μία και ζουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν για αυτές τις επιχειρήσεις από την άλλη. Δυστυχώς τα δικαιώματά τους δεν γίνονται σεβαστά. το, και το λέω με τον ευρύ τρόπο αυτό. Δηλαδή, τα δικαιώματά τους ως άτομα καταρχήν. Ως εργαζόμενοι και ως πολίτες. Η έλλειψη αυτού του σεβασμού οδηγεί σε διαφοροποίησεις. Μπορεί να οδηγήσει σε αθέμητο ανταγωνισμό αυτή η διαφορά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημία ως προς τα άτομα τα οποία δεν ε, από το σεβασμό που θα έπρεπε να είχαν κανονικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό τον, αυτή την ενιαία παλέτα δικαιωμάτων ε, δεν μπορούμε να την ε, βάλουμε στον ίδιο ντουρβά. Και δεν είναι αρμοδιότητα μία και μόνο κοινοβουλευτική επιτροπή. Ένα τρόπο όμω συντονισμού των δράσεων. Ε, Παρ' όλα αυτά θα ήταν χρήσιμο. Δεν πρέπει μία επιτροπή να παίρνει, να έχει την πρωτοκαθεδρία εναντί μια επιτροπη να παιρνει να εχει την καθεδρια εναντι μια αλλη Ε, δεν πρέπει επίση να έχουμε τομεακέ προσεγγίσεις. Όχι, πρέπει να έχουμε σφαιρικέ προσεγγίσεις. Δεν πιστεύετε ότι σε πολλέ δραστηριότητε υπάρχει ένα έλλειμμα προ τα δικαιώματα. Και δεν ξέρω αν στη δουλειά εσεί που κάνετε δεν έχετε ανάγκη να εξασφαλίσετε ένα τόπο, ας πούμε, να, να, να υπάρχει ένας χώρος όπου μπορούμε να διαφυλάξουμε αυτά τα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντικό το ζήτημα που αναφέρατε. Εγώ πρέπει να φύγω στις 4.30 και οι δύο κυρίες που έκαναν τις πρώτες ερωτήσεις θα ήθελαν να παρεύουν και αυτές. Ε, κυρία Κορατσαμπέλτ, να είστε σύντομοι παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την γενναία σα, σας. Μια διευκρίνηση κύριε Υπουργέ όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες εκτιμάται το ενδεχόμενο αύξηση 2,6% αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Εσείς είπατε θα υποστηρίξετε την Κομισιόν στη δουλειά τη. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί η Κομισιόν είπε ότι θα έχει μηδενική ενοχή, αλλά θα ήθελα, αν μπορώ να σα αποσπάσω, μια δέσμευση προ τα κράτη-μέλη, διότι υπάρχει μια ομάδα εργασία για την οδηγία για τις υπηρεσίες όπου ακούγονται πολύ ωραίες διπλωματικές ε, θέσεις, χωρίς να θέλω να κατονομάσω κάποιον. Ελπίζω πραγματικά ότι η Ελληνική Προεδρία θα μπορέσει να πάρει πρωτοβουλίες. Έχουμε τώρα την αξιολόγηση τίμων τη σύνδεση με το εξάμεινο που είναι στα χέρια του Συμβουλίου. Μπορώ να σας αποσπάσω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ και η κυρία Πέντρικα τέλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για άλλη μια φορά θα ήθελα να επαναλάβω τι ευχαριστίες μου προ τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του εδώ στην Επιτροπή μας ε, και θα ήθελα να σας ευχηθώ ότι καλύτερο κατά την καθήκηση των εργασιών του Συμβουλίου κατά την Ιρλανδική Προεδρία. Και δεν συνηθίζουμε να λιθοβολούμε τους υπουργούς μας ε, στην Ιρλανδία, ήθελα να πω. Εμείς ε, προσπαθούμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας και στις επιχειρήσεις μας την ευκαιρία να ζουν, να, κάνουν εμπόριο και να δραστηριοποιούνται χωρίς σημαντικά εμπόδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ιρλανδοί φυσικά γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη μελλοντική μας ευημερία. Εμείς ε, είμαστε δεσμευμένοι για το όλο ευρωπαϊκό έργο από την αρχή και χαίρομαι γι' αυτό, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η διακυβέρνηση στην Ευρώπη θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δουλειά που κάνουμε σε αυτή την Επιτροπή. Διότι η σταδιακή ολοκλήρωση της ε, ενιαίας αγοράς, όπου αυτή τη στιγμή εστιαζόμαστε σε δημοσιονομική λιτότητα, τον αποπληθωρισμό και αυτό Ελπίζω επειδή τα κράτη-μέλη κάνουν κυρίως εμπόριο μεταξύ τους, φοβάμαι μήπως καταλήξουμε σε ε, ένα πολύ ωραίο μηχανισμό ενιαίας αγοράς, ε, ο οποίος δεν θα μπορεί να κινηθεί. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε κύριε ε, Υπουργέ, αλλά η ερώτηση προς εσάς είναι πώς βλέπετε να συνεργάζεστε με τους υπουργούς που είναι επιφορτισμένοι με το ECOFIN και Πού πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσετε. Ε, και εγώ πρόκειται να είμαι τη ηγετρία για το σύστημα ηλεκτρονικών συστημάτων και θα ήθελα να μου πείτε τι προτίθεστε να κάνετε για αυτό το σημαντικό σύστημα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ευχαριστώ και ξανά κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε κυρία Πρέντεργκαστ. Τελευταίες απαντήσεις λοιπόν. θέσατε. Το ζήτημα, κυρία Λεγκρίπ, ε, του τελωνιακού κώδικα. Σίγουρα εμείς ε, προωθούμε τις συζητήσεις, εντατικές συζητήσεις στις ομάδες εργασίας. Αντιλαμβάνομαι το έργο του Κοινοβουλίου γι' αυτό και πράγματι ε, έχετε, στο παρελθόν έχετε παράσχει πολύ αποτελεσματικά μέτρα για την Τελωνιακή Ένωση και αυτό δείχνει πόσο δεσμευμένοι είστε και πόσο συνεργάσιμοι. Αν λοιπόν και εμεί να επιτύχουμε αυτή την προθεσμία, νομίζω ότι είναι 24η Ιουνίου και είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ε, ζητήματα που εκκρεμούν ακόμη και ορισμένα από αυτά είναι αρκετά τεχνικά και δύσκολα. Σίγουρα όμως έχουμε δεσμευτεί να τηρήσουμε αυτή την προθεσμία και βάσει... Οι, οι που έχουμε με τα κράτη-μέλη προχωρούν πολύ καλά και αυτό με ενθαρρύνει Αναφέρατε και κάποια άλλα ζητήματα όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο Συμβούλιο. Εργαζόμαστε για να πλήσουμε ζητήματα όπως η απόσπαση των εργαζομένων, την αφορητότητα των συντάξεων, τα επαγγελματικά προσόντα φυσικά, αποτελεί ζήτημα για τη δική σας επιτροπή. Όλα αυτά είναι κομμάτι αυτής της ισορροπίας, ε, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι εργαζόμενοι δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευση όταν εργάζονται σε άλλα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με αυτό που είπατε. Πρέπει να επιτευχθεί η ισορροπία, η θα είναι πολύ σημαντική για αυτό το ζήτημα, μέσω μια σειρά μέτρων που θα υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλιστεί το άνοιγμα των αγορών και η δίκαιη μεταχείριση. Βρισκόμαστε σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Απασχόλησης και εκεί αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα Εγώ έχω το πλεονέκτημα ότι βλέπω και τις δύο πτυχές του νομίσματος και ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε και στους δύο τομείς. Άκουσα αυτό που είπατε, ότι πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί στην εφαρμογή. Η Προεδρία θέλει να καταγραφεί με πιο ανοιχτό τρόπο η πρόοδος και ξέρω ότι η Προεδρία δεν έχει άλλο ρόλο πέρα από την, το να προεδρεύει. Δεν είμαστε εκτελεστικό όργανο. Ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και φυσικά ε, υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις μέσα στο Συμβούλιο, θα πρέπει να τις συγκεράσει η Προεδρία. Ε, πολύ σωστά εκφράσατε αυτή τη φιλοδοξία, συμφωνώ. Από την άλλη όμως ε, το αξίωμά μας, η Προεδρία μας ε, εμπεριέχει και κάποιους περιορισμούς το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας έχει φιλοδοξίες, θέλει να είναι πιο αυστηρό. Ε, ευχαριστώ τη Φιλίπα για τα ευγενικά της σχόλια στην πρώτη παρέμβαση και τα τελευταία της σχόλια. Φιλίπα, έθεσε ένα σημαντικό ερώτημα για την ισορροπία και τη στρατηγική ε, διόρθωσης Θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η στρατηγική ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντική, πέρα από την δημοσιονομική πτυχή. Φέτος υπάρχει μια αλλαγή στην προσέγγιση, ε, καταγράφεται στο εξάμεινο και η Επιτροπή Απασχόλησης και το ΕΠΣΚΟ θα έχει σημαντικότερο ρόλο στην όλη διαδικασία θα σκεφτούμε χωριστά τα θέματα που αφορούν την απασχόληση και απασχολούν τους υπουργούς απασχόλησης. Και στο ΕΠΣΚΟ και στο ΕΚΟΦΗΝ θα ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά, ούτω ώστε και οι δύο απόψεις να λυθούν υπόψη. Και στο ΕΠΣΚΟ και στο ΕΚΟΦΗΝ. Δεν υπάρχει ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή, η δημοσιονομική εξυγίανση είναι εκ των όνου Αλλά χρειαζόμαστε επίσης ε, εργαλεία για να δημιουργηθούν ευκαιρίες, επενδυτικές, που να μην βασίζονται όμως ε, στα δημοσιονομικά ελλείμματα. Χρειαζόμαστε στρατηγικές για να ανοίξουμε το εμπόριο. Αυτές οι στρατηγικές πρέπει να προωθηθούν και να διορθώσουμε βεβαίως και τις αποτυχίες της αγοράς. Γιατί πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν προβλήματα με τις τράπεζες. Ε, προφανώς η αγορά δεν βρίσκεται στο ύψος των προσδοκιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχουν μια πλειάδα παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν εκ παραλλήλου. Αυτή την ισορροπία προσπαθούμε να επιτύχουμε. Βεβαίω θα κάνουμε πολιτικά παζαρέματα για να δούμε πού θα πετύχουμε αυτή την ισορροπία, αλλά η Προεδρία θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της μια ευρία, ένα ευρύ φάσμα πούμε, εργαλείων αν θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή ανάπτυξη. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Όπως είπα και στην αρχή, το εντυπωσιακό με την ε, Ιρλανδική Προεδρία είναι ότι εσύ, Ρίτσαρντ, και οι συναδελφοί σου ξέρετε πολύ καλά τα θέματά σα και τα απεικονίζετε με πολύ καλό τρόπο. Όπω είπε προηγουμένω, Ρίτσαρντ, η δουλειά μα είναι να προσπαθήσουμε να δώσουμε κίνητρα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ξέρουμε ποιο είναι ο ρόλο μα, αλλά θέλουμε να προωθήσουμε και κάποιε μακροπρόθεσμε μεταρρυθμίσει, αμοιβαία αναγνώριση, δημόσιε προμήθειε Γι' αυτό βασιζόμαστε στην υποστήριξή σα. Θα είναι κρίσιμη αυτή η περίοδο. Θα προσπαθήσουμε αυτό το διάστημα να δώσουμε αποτελέσματα. Πολλοί από τους ε, εισηγητέ και σκιώδει εισηγητέ είναι εδώ. Ε, Ρίτσαρτ, ε, περιμένω να σε ξαναδώ. Και στο μεταξύ θα συναντηθούμε και εκτός συνεδριάσεων της Επιτροπής. Ούτως ή άλλως από την ε, ιδιαίτερη πατρίδα μου στο Δουβλίνο ε, μπορεί κανείς να πετάξει σε ένα πολύ μικρό διάστημα. Ελπίζω λοιπόν να τα ξαναπούμε και φαντάζομαι ότι πολλοί από τους βουλευτές συμφωνούν με αυτά που είπα. Ah, you can have the floor later. It's to congratulate you personally. But uh, so, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, τώρα είμαστε στο τελευταίο θέμα γιατί μετά έχουμε συντονιστές. Στόχος μας είναι να συζητήσουμε δημόσια πριν ψηφίσουμε αύριο. Μετά το μαραθώνιο έργο του Μάρκ Ταραβέλα που έχει να κάνει με τις συμβάσεις σε τομείς υπηρεσιών κοινή ωφελία. Το συζητήσαμε και πριν τα Χριστούγεννα, είμαστε στα μέσα του δρόμου δηλαδή. Αύριο είπαμε θα ψηφίσουμε. Συνεπώς, τώρα χαίρομαι πάρα πολύ που είναι εδώ ο κύριος Ταραμπέλα. Έχουμε και δύο σκιώδεις, τον κύριο Έγκελ και εγώ ίδιος είμαι εδώ. Α, κυρία Ρούλε, τρεις σκιώδεις είμαστε εδώ. Τους φιλελεύθερου δεν έχουμε. Ο κύριος Κρότσμαν είναι εδώ. Όχι. Μπορεί να έρθει αργότερα. Στο μεταξύ θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας για να μας πει πού βρισκόμαστε όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες ή οτιδήποτε άλλο θέλει να μας πει. Εν πάση περιπτώσει να ψηφίσουμε αύριο στην Επιτροπή μας. Κύριε Ταραμπέλα, έχετε το λόγο. Merci, euh, cher président, cher Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα ήταν λιγότερο δύσκολα τώρα από την προηγούμενη φορά, γιατί πρόκειται για το δεύτερο τμήμα αυτή τη ειδική οδηγία. Πρόκειται, όπω είπαμε, για το ίδιο την ενέργεια, τι μεταφορέ και τι ταχυδρομικέ υπηρεσίε, για του αφηρημένου το λέω. Τα δύο κείμενα βέβαια μοιάζουν, πράγμα που σημαίνει ότι μπορέσαμε να δουλέψουμε με συνοχή και έτσι να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές προτάσεις όσον αφορά τις τμηματικές οδηγίες σε σχέση με τη συνολική οδηγία του Δεκεμβρίου και πέρα από δύο συμβαστικέ προτάσεις για δύο τελογικές σκέψει. κατά τα άλλα υπήρξαν 89 συμβαστικέ από τι 91 που προτάθηκαν, 89 έγιναν αποδεκτές. Με ευρία, με λιγότερο ευρία πλειοψηφία, με πλειοψηφία πάντως. Στην Επιτροπή μας στις 18 Δεκεμβρίου. Τα κείμενα βέβαια διαφέρουν κάπως. Έχουν να κάνουν ιδιαίτερους τομείς και έτσι προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερους συμβιβασμούς να δεχτούμε. Ε, θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε τις συμβαστικές προτάσεις όλες μαζί, αλλά επειδή δεν είναι τόσο φοβερό, θα έλεγα μία-μία τις συμβαστικές προτάσεις να τις ψηφίσουμε. Τώρα, συνήθως είμαι πολύ ανοιχτός, σαν στρίδι, ανοίγω εύκολα, αλλά μερικές φορές κλείνω κιόλα. Και θέλω να πω σε όσους θέλανε να προσθέσουν ε, προτάσεις κτλ. Και, και εγώ θα ήθελα. Δεν το έκανα όμως. Και αυτό γιατί νομίζω ότι η ψηφοφορία ήταν σαφής και καλό είναι να μείνουμε εκεί και να μην ξανανοίξουμε χωρίς λόγο τη συζήτηση. Σας λέω και εγώ θα ήθελα να προτείνω και άλλες αλλαγές. Δεν το έκανα όμως. Συγκρατήθηκα. Γι' αυτό και δεν θα ήθελα να ξανανοίξει η συζήτηση. Και ο Έγγελ νομίζω ότι συμφωνεί. Υπάρχουν όμως τέσσερα σημεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ, στα σημεία 27 και 28, τα οποία έχουν να κάνουν με δραστηριότητες οι οποίες είναι αντιμέτωπες με τον ανταγωνισμό. Το άρθρο 11 που είναι η τροπολογία με 25 που αναφέρεται στις εξαιρέσεις τμήματων υπάρχουν κάποια άρθρα για τα οποία δεν καταλήξαμε σε συμβιβασμό. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε τροπολογίες που δεν θέλουν να αποκλείσουν τομεί σε κάποιους συγκεκριμένους τομεί. Και στο άρθρο 27, όταν μία δραστηριότητα είναι αντιμέτωπη με τον ανταγωνισμό, τότε η υπηρεσία, ο φορέας μάλλον, ο οποίος ε, αποφασίζει για τις δημόσιες ε, ε, συμβάσεις, μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την οδηγία, και αυτό λέει και το άρθρο 28 οι 431, 433, 435, 436, 438, 440 και 442 Αντσελίκ, Τιρνενστάιν, Σακτρακόφσκι και οι τροπολογίες 432, 434, 437, 439, 441, 443 και 444 Κόμνου Μπαλτασάρε νομίζω ότι πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση όμως δεν λύνουν το πρόβλημα για το πώς θα προχωρήσει η εμπορική στρατηγική. Γι' αυτό θα ήθελα να στηρίξουμε στο άρθρο 11 τη δικιά μου τροπολογία 25. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ταχυδρομεία. Ξέρω ότι ορισμένα ταχυδρομεία θέλουν να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Το αρνήθηκα πάντα, διότι αποτελούν μέρος των κοινοφελών αυτών υπηρεσιών. Αν μέρη είναι ιδιωτικοποιημένες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάποια υπηρεσία που συνήθως προσφέρει το κράτος. Όταν όμως το ταχυδρομείο υποβάλλεται σε κάποιο τμήμα της δραστηριότητάς του στον ανταγωνισμό με επιχειρήσεις καθαρά ιδιωτικέ που πάντα ήταν ιδιωτικέ, το UPS για παράδειγμα, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά ε, πάει και μοιράζει τα δέματα στα σπίτια. Τότε, λοιπόν, άμα θέλει να αγοράσει ένα ε, φορτηγάκι για να μοιράζει τα πακέτα, θα άνοιγε την στρατηγική της, την εμπορική προς τα έξω. Και εκεί ε, έχει να κάνει η τροπολογία με 25. Το ίδιο και για την 22 που έχει να κάνει με τις συνδεδεμένες υπηρεσίες. Αυτό το άρθρο αποτέλεσε αντικείμενο συμβιβασμού αλλά με και έναν παραλυσμό με τις παραχωρήσεις, γιατί την ίδια έννοια τη βρίσκουμε και στην οδηγία για τις παραχωρήσεις. Ο κ. Ζουβάν είναι ο συγητής. Τα είπαμε μεταξύ μας. Θελήσαμε να έχουμε μια συνοχή, οπότε η συμβαστική λύση είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο σημείο, άρθρο 82, στις ε, εναλλακτικές, τις παραλλαγές. Και εδώ πάλι δείξαμε ευαισθησία στους τομείς όπου εφαρμόζεται και είπαμε να υπάρξει κάποια ελαστικότητα για να μπορούμε να προβλέψουμε ένα περιθώριο ελιγμών σε περίπτωση που υπάρχει κάτι που καθυστερεί ένα εργοτάξιο, να μην δαπανώνται χωρίς λόγο χρήματα. είναι λογική δηλαδή θεωρήσαμε ότι είναι η ελαστικότητα. Και όσο για το παράρτημα 3, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στην ε, μεταφορά εμπορευμάτων ότι εξαιρείται από την οδηγία δεδομένου ότι εκτίθεται στον ανταγωνισμό η υπηρεσία αυτή βάσει τη 91440. Σύμφωνα με τα τελευταία που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ολοκλήρωση της αγοράς 2013, οι επιβατικές μεταφορές από το 2010 είναι ανοιχτές στον ανταγωνισμό. Οπότε η ίδια οδηγία ανοίγει τη μεταφορά εμπορευμάτων ε, με τρένο και τις επιβατικές συγχρόνως. Αυτά είναι στο παράρτημα 3. Τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι δουλέψαμε μέσα σε ένα εξαιρετικό πνεύμα. Νομίζω ότι τα δείγματα που έχουμε είναι θετικά για τις διαπραγματεύσεις. Σήμερα το πρωί είδα τον Ιρλανδό Υπουργό προγευματίσαμε μαζί. Δεν αρχίσαμε διαπραγματεύσεις, ήταν απλώς μια επαφή που είχαμε. Και δείχνει και αυτός ότι το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να προχωρήσουμε και να καταλήξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε αυτή την υπόθεση. Ελπίζω ότι θα βρούμε την καταλληλότερη διατύπωση έτσι ώστε να έχουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μπορέσουμε να επιμείνουμε σε αυτήν Για να την περάσουμε. Αυτό θέλουμε, από την αρχή το θέλαμε. Γι' αυτό και θα συζητήσουμε επί της διαδικασίας αργότερα, ίσως όχι τώρα. Εγώ προτείνω μια μέθοδο που να μας οδηγήσει στον τριμερή διάλογο όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εντάξει, δεν θα το αποφασίσω εγώ σήμερα, θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις. Πάντως, ο καρπός είναι όριμος και πρέπει να τον μαζέψουμε, Πρόεδρε. Μην τον αφήνουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνοπτική αυτή παρουσίαση. Τονίσατε τις σημαντικές διαφορές και ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια που αντικατοπτρίζονται καλύτερα στις συμβαστικές που εξετάζουμε. Ε, ας ακούσουμε τα σχόλια των σκιωδών, ξεκινώντας από τον κύριο Έγκλ, τον κύριο Κρότσμαν, την κυρία Ρούδερ και μετά η, θα να... η κυρία Γκέπχαρτ θα ήθελε να μιλήσει. Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Έγκρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος. Πρώτα απ' όλα ο εισηγητής, ο συνάδελφος και φίλος κύριος Ταραμπέλα τα είπε ουσιαστικά όλα. Ό,τι υπάρχει να υποθεί σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο για την αυριανή ψηφοφορία που ευθυγραμμίζεται στο βαθμό που ήταν δυνατόν σε ό,τι ψηφίσαμε τον Ιανουάριο, τη μεγάλη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο είναι λογικό. Αυτή μας επέτρεψε να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα και β' αρκετά άνετα, ουσιαστικά στην ίδια βάση, όπως το παρελθόν. κάποια πράγματα δεν ήταν δυνατά παρότι κάποια λόμπι τα επιθυμούσαν πολύ. Έτσι έχει η ζωή. Τι να κάνουμε. Το να μην εξαιρείται αύριο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες από κάθε εφαρμογή ήταν κάτι για το οποίο δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι στα όσα είπε ο κύριος Ταραμπέλα για αυτό το θέμα. Όσον αφορά διαδικασία, Αύριο θα συζητήσουμε μετά την ψηφοφορία, όπως έχει συμφωνηθεί, στις συμφωνημένες βάσεις, όπως ορίστηκα μετά από αυτές τις δύο μεγάλες ψηφοφορίες, λοιπόν, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Δεν θα ήθελα να πω ψέματα σε όσους ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, με αυτό το φάκελο σε αυτή την αίθουσα. Όλοι μας έχουμε λίγο κουραστεί και θα θέλαμε, ακόμη και αν δεν είναι πολύ εύκολα, να έχουμε τελειώσει μέχρι το Πάσχα. Ευχαριστώ. Και εγώ το ίδιο επιθυμώ. Επιθυμούμε όταν θα βγουν τα λούδια την άνοιξη να ανθίσει και αυτή η νέα οδηγία. Κύριε Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον κύριο Συγητή του Σκιώδης και τη Γραμματεία. Σε πολλούς από αυτούς τους τομείς, όπως είπε ο κύριος Ταραμπέλα, καταφέραμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβιβασμούς και σε συμφωνίες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Όπως είπε ο κύριος Ταραμπέλα, συνδέονται όλα αυτά με τις εργασίες μας στο παρελθόν. έχουμε τα ίδια προβλήματα να αντιμετωπίσουμε όπως είχαμε και τότε. Όσον αφορά τις τομεακές οδηγίες υπάρχουν προβλήματα. Η ευθύνη των ε, υπεργολάβων είναι ένα τομέα ε, και εργαζόμαστε. Φαίνεται σαν να μην θέλουμε να υποστηρίξουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά δεν είναι αυτό αλήθεια. Απλά προσπαθούμε να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Η πρόταση της Κομισιόν θεωρήσαμε εμείς θα ήταν καλύτερη. Διαφορετική. Αλλά καλύτερη. Τώρα ο κύριος Ταραμπέλα είπε ότι θέλει να περάσει αμέσως σε ψηφοφορία, σε δοκιμαστική ψηφοφορία, γιατί σε, συγγνώμη, σε τριμερή διάλογο. Αλλά είναι αυτή η καλύτερη ιδέα, γιατί αν πούμε κατευθείαν σε τριμερή διάλογο, αυτό θα λειτουργήσει. Θα λειτουργούσε μόνο αν είχαμε τρει-τέσσερι ψήφου κατά και δύο-τρει αποχέ. Αλλά αν αυτό δεν συμβαίνει, αν δεν υπάρχει τέτοια καθαρή γραμμή, κύριε Ταραμπέλα, τότε όσοι είναι υπέρ και ο Μάρκολμ Χάρμπορ το γνωρίζει, Είχα εγώ το ίδιο πρόβλημα με τον τριμερή διαλόγο για τα πνευματικά δικαιώματα. Χρειάστηκε να αναφέρομαι ξανά και ξανά σε μια κοινοβουλευτική απόφαση και υπήρχε μια περίπτωση όπου υποστηρίζαμε την Κομισιόν αλλά η Ολομέλεια είπε δεν τα θέλουμε όλα αυτά και το Συμβούλιο είπε το ίδιο. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτή ήταν η άποψη της Ολομέλειας. Θα μπορούσα να το είχα διαπραγματευτεί διαφορετικά στον τριμερή διάλογο. Αν είχα πει ότι αυτό θέλει η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και ο Μάλκομ συμφωνούσε με μαζί μας θα ήταν καλό το αποτέλεσμα. Αλλά όταν η ψηφοφορία είναι επίμαχη σε μια ε, αντιφατική σε μια επιτροπή και δεν θέλει κανείς να είναι το ίδιο στην Ολομέλεια, χρειάζεται κανείς να ενισχύσει τη θέση του. Ο συζητητής και με τον πρόεδρο μαζί μου είχαμε δυσκολίες και αποφασίσαμε ότι στο μέλλον, στις Ολομελίες, θα κάνουμε τα πάντα σε πρώτη ανάγνωση. Μου έκανε έκπληξη. Πότε ξεκινάει το μέλλον. Μετά τις επόμενες ευρωεκλογέ, αναρωτιέμαι, τότε ξεκινάει το μέλλον. Πότε πρόκειται να ξεκινήσει αυτό το μέλλον ή είναι να ξεκινήσει τώρα. Αυτά είναι τα σχόλια που ήθελα να κάνω, διότι ο κύριος Ταραμπέλα με τον οποίο έχω εξαιρετική εργασιακή σχέση θέλει να στρωθεί στη δουλειά ευθύ αμέσω. Γνωρίζω ότι και η Επιτροπή θέλει να στρωθεί στη δουλειά γι' αυτό, αλλά αναρωτιέμαι για ποιο λόγο θέλει τόσο πολύ η Επιτροπή κάτι τέτοιο. Το θέλει διότι Πιστεύετε ότι το Συμβούλιο συμφωνεί ότι μπορούμε να περάσουμε απευθεία σε τριμερή διάλογο και να κάνουμε τα πράγματα γρήγορα. Ταυτόχρονα είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή έχει κάποιους καλούς λόγους για να θέλει να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο. Ευχαριστούμε που προετοιμάζετε έτσι τη συζήτηση. Θα είμαι σύντομος και πρακτικός. Προσπαθώ να παραμείνω ουδέτερο επί του θέματος. Αυτή είναι η δουλειά μου ως πρόεδρος. Κύριε Αβέλα. Ευχαριστώ. Δεν είναι τίποτα ουδέτερο. Και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Κρότσμαν και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Και ζητάω από τον εισηγητή να θυμηθεί αυτό που έχουμε πει κατά το παρελθόν. Οι, οι είχαν πάντα πει ότι σε αυτό το θέμα είτε ότι πρέπει να σεβόμαστε τις δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι καλύτερα να θεωρήσουμε ότι είναι σε αυτήν ε, την κατηγορία τη στιγμή που ξέρουμε ότι έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ να οφείλεται στις δημόσιες συμβάσεις. Στον τομέα αυτό λοιπόν επίγει να ενισχύσουμε τους δημοκρατικούς, τις δημοκρατικές αρχές. Εφόσον ψηφίσαμε όπως ψηφίσαμε, δεν μπορούμε να έχουμε τώρα αντίλογο, θα έλεγα, να το θυμόμαστε και να θυμόμαστε τι έχουμε πει κατά το παρελθόν για, τα, για τέτοιου είδους θέματα. Ο κύριος Κρότσμαν έχει δίκιο. Αυτός θα πρέπει να είναι ο κανόνας στο μέλλον. Αυτό λοιπόν πιστεύω εγώ τώρα για αυτά που είπε ο κύριος Ταραβέλα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν τρεις ομάδες οι οποίες δεν ανέκριναν την έκθεσή του, δεν συμφωνούν μαζί του. Και υποθέτω ότι ούτε και αύριο θα αντιστηρίξουμε την έκθεση αυτή. Εμεί θα κρατήσουμε θέση αποχή πάντω, όπω κάναμε και την προηγούμενη φορά και για του ίδιου μάλιστα λόγου. Ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δεν συμφωνούμε με τον τρόπο αυτό που αποφασίζουμε για τι δημόσιε συμβάσει, την αμοιβαιότητα, ούτε συμφωνούμε με την υπεργολαβία δεν έχουμε την ίδια απόψη με εσά, κύριε Ταραμπέλα. Και έχω την εντύπωση ότι καλό θα ήταν να συζητήσουμε εκτενώς το Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Ως εισηγητής θα έπρεπε να ε, συμμορφωθείτε προς τη συζήτηση που θα κάνουμε και μετά έτσι να πάτε στον τριμερή διάλογο. Είναι κρίμα για σας τώρα το να πάτε εκεί και να υποστηρίζετε πράγματα με τα οποία δεν συμφωνείτε. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο για εσάς. Πρόεδρος, Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Για να το ξεκαθαρίσω. Ως και ο συζητητής θα σας πω ότι και εμείς κρατήσαμε την τελευταία φορά αποχή, θέση αποχής. Συνεισφέραμε στη διαδικασία, προσπαθήσαμε και εμείς να συνεισφέρουμε στις συμβαστικές τροπολογίες, αλλά τα πράγματα έχουν όπως έχουν. Και δεν θα είναι έκπληξη ότι είμαστε κατά της ε, αμεβαιότητας και την προηγούμενη φορά, όπως επίσης και για την υπεργολαβία. Δεν θα επαναλάβω τώρα τα επιχειρήματά μου γιατί είμαστε κατά. Με τον ε, σωστό τρόπο πρέπει να χειριστούμε αυτά τα θέματα, είναι αλήθεια. Το πρόβλημα δεν είναι ο χειρισμός τους, το θέμα είναι ότι πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος να τα χειριστούμε. καταφέραμε να προχωρήσουμε κρατώντας κάποια συνοχή με την οδηγία για να αντικατοπτρίζονται οι διαφορές μας όσον αφορά τις συμβάσεις για αυτές τις υπηρεσίες που εξετάζουμε εδώ. Όντως υπάρχουν ιδιαιτερότητες και στις δομές των συμβάσεων. Το έχουμε δει αυτό από την οδηγία για τις κοινοφελή αυτές υπηρεσίε. Τώρα το επόμενο στάδιο, στο επόμενο στάδιο πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου. Γιατί αν είναι να μπούμε σε διαπραγματεύσεις πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει βούληση για διαπραγμάτευση από την άλλη πλευρά. Ο υπουργό αυτό μας είπε. Παρ' όλα αυτά θα έπρεπε να έχουμε κάποιο κείμενο από αυτούς, επίσημο είναι, φαίνεται άκρος απόρριτο. Δεν το έχουμε. Η κρίσιμη απόφαση για τα μέλη της Επιτροπής μας, και εδώ σας μιλάω ως πρόεδρος και πάλι, και όχι ως Σκιώδης, γιατί εγώ θα πρέπει να ακολουθήσω αυτά που θα μου πείτε στις διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, η κρίσιμη απόφαση θα είναι πώς θα ευθυγραμμίσουμε τη δικιά μας τη θέση με εκείνη του Συμβουλίου που κάποια στιγμή θα δημοσιοποιηθεί βέβαια. Και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να μείνουμε στην θέση του Κοινοβουλίου. Γιατί η βασική πολιτική κατεύθυνση του Συμβουλίου είναι γνωστή. Αυτά λοιπόν είναι τα επίμαχα. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε βελτίωση για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δημόσιες συμβάσεις. Είναι καλό για την οικονομία, για τις μικρές επιχειρήσεις, για το περιβάλλον, διότι έχουμε πιο πράσινες λύσεις, έτσι. Και θα είναι και καλό για όλους όσοι απασχολούνται στα θέματα αυτά. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικά. Σημαντικά επιτεύγματα. Πότε όμως θα τα καταφέρουμε, πότε θα τα γιατί όπως είπε και η κυρία Ρούλε, δεν μπορεί να είναι μυστικά. Θα θυμόσαστε ότι στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών είχαμε κάπως διαφορετική θέση όταν αρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις και η θέση του Συμβουλίου ήταν πολύ μακριά από τη δικιά μας. Θα το θυμάται ο κύριος Βαπ. Όμως, συνδυάσαμε τα πράγματα, αρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, σιγά σιγά πιέσαμε και τελικά ψηφίσαμε. Σας υπενθυμίζω ότι αν ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, τότε ο χρόνος που έχουμε για διαπραγμάτευση μετά περιορίζεται. Πέντε εβδομάδες, έτσι δεν είναι. Το κοιτάω κι εγώ εδώ πέρα με τον ε, τμήματάρχη μου. Μερικές φορές είναι πολύ σημαντικό να πιέζουμε με το χρόνο για να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Δεν θα ήθελα βέβαια να διακινδυνεύσουμε την ποιότητα. Ποιότητα και χρόνος είναι δύο παράγοντες που πρέπει να τους σταθμίσουμε καλά και ισορροπημένα. Άκουσα αυτό που είπε η κυρία Ρούλε. Ας κάνουμε πρώτα ένα προκαταρτικό γύρο συζητήσεων να δούμε πού, πόσο ευθυγραμμίζονται οι θέσεις μας και μετά να αποφασίσουμε. Σας είπα τις σκέψεις μου, χωρίς να κάνω σύσταση. Έχει προχωρήσει πάντως οι θέσεις μας πολύ. Αύριο θα είναι κρίσιμη η στιγμή για την ψηφοφορία. Στην πράξη, μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάτι το δεν μου φαίνεται ρεαλιστικό, αλλά μπορούμε ίσως να προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Δεδομένης όμως της δουλειά που είχαμε και τις τροπολογίες, αυτό δείχνει ότι αν μη τι άλλο είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και να δουλέψουμε σκληρά. Καλό ήταν αυτό. Κυρία Κέπαρτ, άλλος κανείς. Αν κάποιο κοιόδη ηγητή θέλει να ξαναπάρει το λόγο, ε, θα τον δώσω. Αλλά α ακούσουμε την κυρία Γκέπχαρτ, ο κύριο Έγκχαρτ και ο κύριο Κρόιτσμαν, ο κύριο Φαμπ. Κυρία Ρούλε. Όλοι θέλουν ξανά το λόγο. <laughs> Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω τη συζήτηση που κάναμε σήμερα το πρωί, αλλά θέλω να σας πω το εξή. Η ομάδα μου αύριο θα έχει σκεφτεί για τη διαδικασία. Όλοι εξαρτώνται από το αποτέλεσμα ψηφοφορίας. Ε, και αυτό θα, το αποτέλεσμα ψηφοφορίας θα καθορίσει τη θέση μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να πω σήμερα τι θα κάνουμε και τι δεν θα κάνουμε. Κυρία Ρούλε, σας υπενθυμίζω ότι δεν έχει νόημα να υποστηρίζουμε εδώ στην Επιτροπή κάποια πράγματα που δεν υποστηρίζουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Εσείς, κυρία Ρούλε, δεν πήρατε το λόγο να τοποθετηθείτε σε αυτά που σας είπα στις συνεδρίες των συντονιστών. Τέλος πάντων, θέλω να ευχαριστήσω τον Μάρκα Ταραμπέλα, τον κύριο Έγγελ, Έγγελ και όχι Έγγελς, Κύριε Έγγελ, ζητώ συγγνώμη που σας μπέρδεψα με κάποιον με τον οποίο δεν έχετε καμία σχέση. Τέλος πάντων, Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη θαυμάσια συνεργασία που είχαμε. Δεν ήταν πάντα εύκολα τα πράγματα. Δεν ήταν πάντα εύκολο γιατί χρειάστηκε να κάνουμε όλοι μας προσπάθειες να δεχθούμε να κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς. για να υπάρξει μια κοινή θέση στην Επιτροπή είναι, ήταν εφικτό για πολλά δύσκολα θέματα αυτό και αυτό ήταν θαυμάσιο. Οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι άσκησαν ε, κριτική για ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μας. Τα κοινωνικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην διαδικασία ανάθεσης. Αυτές οι αρχές θα πρέπει να λαμβάνονται όχι μόνο υπόψη, όχι μόνο από τον ανάδοχο, αλλά και από τους υπεργολάβους. Αυτό για μας είναι απαραίτητο. Τι νόημα έχει να γίνονται σεβαστά αυτά τα κριτήρια από τον ανάδοχο, αλλά όχι από τους υπεργολάβους. Αυτό είναι ένα από τα σημεία που υπάρχει στην έκθεση του Μάρκ Ταραμπέλα και μου επιτρέπει να πω ότι πετύχαμε ένα καλό συμβιβασμό, συμβιβασμό. Ακούγονται διάφορα εκτός μικροφώνου. Ναι, κυρία Γκέπχαρτ, ναι, κυρία Γκέπχαρτ μου. Διάβασα το ανακοινωθέν τύπου σας, αλλά πρέπει να είσαστε πιο ειλικρινείς για αυτά τα θέματα, κυρία Γκέπχαρτ. Μην ξεχνάτε ποιος παρακόλλησε τις ε, διαπραγματεύσεις. Ξέρω πολύ καλά πώς εξελίχθηκαν οι διαπραγματεύσεις που υπήρξαν τα κολλήματα. Τέλο πάντων, τελικά μπορούμε να πούμε ομως ότι έγινε μια καλή δουλειά. Οι σοσιαλιστες παντως θα στηρίξουν το συμβασμό που έχει επιτευχθεί. Αυτό μπορώ να το πω τελικά. Είναι σημαντικό. και αν υιοθετηθεί ο συμβιβασμό, θα συμφωνήσουμε και με τι διαπραγματεύσει. Για τη διαδικασία θα τα συζητήσουμε μετά. Κύριε Σβάμπ, να μην κάνουμε τώρα την ε, συναντήση των συντονιστών καλύτερα. Τι με νοιάζει εμένα. Απλά ήθελα να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο, διότι νομίζω ότι αύριο θα συναντηθούμε και κλεισμένο των θυρών και αυτή εδώ είναι δημόσια συνεδρία, συνεπώ θα πρέπει να υπάρχει κάτι, να δηλωθεί κάτι δημόσια. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν είμαι βέβαιος για το τι σκέφτομαι για όλα αυτά. Φυσικά Διάβασα την έκκληση που ο Συμβουλίο που πέρυσι ήθελε προσαρμογή αυτής της οδηγίας και η αλήθεια είναι ότι έχουμε δουλέψει πολύ αργά. Θα πρέπει σίγουρα να επιταχύνουμε, πιστεύω θα ήταν καλό. Αλλά όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν επίσης ότι στη ΕΛΚΑ πάντα κρατάμε μια θέση ε, ανοιχτή ως προς την ανάγνωση, ως προς την τοποθέτηση σε πρώτη ανάγνωση και σήμερα διαπιστώνω ότι για αυτή την οδηγία τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Εγώ είμαι ανοιχτό σε όλα, εν τέλει. Αυτό που θα επιθυμούσα, αν ε, εμείς αποφασίσουμε να ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία, προτείνει ο Πρόεδρος, καλό θα ήταν να επιτύχουμε μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Ε, Τίδε διάφορα θέματα, απολύτω εύλογα, που αναφέρουν οι φιλελεύθεροι και όλοι οι υπόλοιποι, θα πρέπει να ενσωματωθούν στο κείμενο. Καλό θα ήταν Λοιπόν, αύριο μετά την ψηφοφορία να μας προβληματίσουν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Πράγματι, η ανάλυση μας έδειξε ότι η απευθεία μετάβαση στην Ολομέλεια προκαλεί διάφορε, ε, σε πολλέ συζητήσει, αλλά όχι πολλέ τροποποιήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι μα συμφέρει να βρούμε μια ρεαλιστική λύση που θα τηρεί τι αποφάσει που λάβαμε και στην Ολομέλεια πριν τα Χριστούγεννα. Ε, άτυπες λοιπόν συζητήσει με την Προεδρία και βάσει όλων αυτών να πάμε στην Ολομέλεια. Αυτό είναι μια λύση που εμένα μου αρέσει, αλλά θα χρειαστεί να το συζητήσουμε και αύριο μετά την ψηφοφορία. Um, Κύριε Κοράτσα Μπίλτη, θέλω να πει δύο λόγια. Ναι, και εγώ θα είμαι γρήγορη. Εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο του Μάρτιν ε, σε αυτό το πολύ δύσκολο ζήτημα. Όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, θα ήθελα να μιλήσω για τη συνοχή. Εδώ δημιουργούμε μια νομοθεσία που χρειάζεται νομική βεβαιότητα για κάποιον που εργάζεται σε έναν δήμο, σε ένα μέρος με ελάχιστους κατοίκους και όταν εκεί χρειάζεται να γίνει εφαρμογή πρέπει να είναι ευκολότερο, πιο απλό, πιο αποτελεσματικό, πιο λογική η νομοθεσία αυτή αφενός. Αυτό, σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Και μετά προσθέτουμε ένα κριτήριο και μετά ένα άλλο ένα και μετά αμέτρητα κριτήρια τα οποία είναι ασαφή. Διότι δεν μιλάμε για κοινωνικά ζητήματα, είναι πολύ δύσκολο να το ορίσει κανείς ποσοτικά. Και ε, τέσσερις φορές αναφέρονται αυτά τα κριτήρια μέσα στο κείμενο και η εφαρμογή καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη και μετά πηγαίνουμε και λέμε ότι θέλουμε να ανοιχτούμε στι μικρομεσαίες επιχειρήσει, να μην έχουν πρόσβαση στη δημόσια συμβάση μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις, ειδικότερα όσον αφορά τι κοινωνικέ υπηρεσίε, τα τρόφιμα και ούτω καθεξής. Και μετά πάμε και προσθέτουμε κριτήρια με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουμε την πρόσβαση των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιε συμβάσεις. Ήθελα λοιπόν από στους φίλου μα να δείξουμε κάποια συνοχή. Μιλάμε για νομοθεσία η οποία πρέπει να είναι υλοποιήσιμη θα πρέπει να εφαρμοστεί σε μικρούς δήμου, σε μικρές κοινότητες και να προσφέρει πρόσβαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσει. Πρέπει να είναι πιο απλή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να προσθέτουμε το ένα κριτήριο μετά από το άλλο. Σε ζητήματα όπως η εργασιακή, οι νόμοι ε, για τους εργαζομένους, για παράδειγμα, που ήδη προβλέπονται στις εργασιακές νομοθεσίες των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, ναι, θα Νομίζω οι σκιώδεις θέλαν να πούνε ένα τελευταίο λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Τραμπέλα. Να ακούσουμε, δεν σας πειράζει να ακούσουμε δύο φορές τους σκιώδεις πριν περάσουμε σε εσάς ξανά. Το έχετε συνηθίσει τους ή άλλως. Λοιπόν, Φρανκ Έγκλ, μπορείτε να μιλήσετε. Κύριε Πρόεδρε, σε δύο πράγματα ήθελα να αναφερθώ. Δεν θα μιλήσω, ήθελα να μην μιλήσω για το κοινωνικό ζήτημα, αλλά όπως φαίνεται δεν γίνεται, δεδομένου των περιστάσεων. Και μετά θα πω δύο λόγια για την αμοιβαιότητα. Ή μάλλον το πω αντίστροφα. Αντίστροφα θα ξεκινήσω από την αμοιβαιότητα. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι θεωρούν ότι συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό το κείμενο λόγια σχετικά με την αμοιβαιότητα αποδυναμώνουμε την ελεύθερες, τις ελεύθερες συναλλαγές. Εγώ θα σας πω πρώτον δεν αληθεύει κάτι τέτοιο. Δεύτερον και η Κομισιόν το είχε προβλέψει στο σχέδιο οδηγίας που ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε αύριο. Δεν κάνουμε λοιπόν κάτι εξαιρετικό σε σχέση με τα όσα είχε ήδη προβλέψει η Κομισιόν παρότι δεν είχε προβλέψει δεν το είχε προβλέψει στο Γενικό Σχέδιο Οδηγία. Μου φαίνεται ότι το Συμβούλιο δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένο. Μου φαίνεται λοιπόν ότι το αποτέλεσμα πριν περάσουμε στην Ολομέλεια θα είναι λιγάκι διαφορετικό από αυτό που κάνουμε ήδη στην Επιτροπή. Αλλά επιμένω. Έχει νόημα να πούμε ότι δεν είναι φυσιολογικό στην Ευρώπη η αγορά μας να είναι ανοιχτή σε όλες και σε όλους, μόνιμα και πουθενά άλλου στον κόσμο δεν μπορούν να έχουν τόσο ελεύθερη πρόσβαση οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει σε καμία αγορά. Δεν υπάρχει λόγο να εξαναγκάσουμε άνοιγμα των αγορών άλλων. Είναι ένα τρόπο να πούμε σε όσους ε, υπάρχουν με του οποίου διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή τις συνθήκε πρόσβαση στην αγορά, να του πούμε ότι πραγματικά επιθυμούμε να ανοίξουμε την αγορά, ώστε και οι υπόλοιποι να κάνουν το ίδιο. Και ότι όσοι δεν πράξουν το ίδιο, στο μέλλον θα τους αξιολογήσουμε κατά περίπτωση, κατά πόσο θα επιτρέψουμε σε μη ευρωπαϊκέ επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Όλα αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. ούτω ή άλλω. Ε, έχουμε συμπεριλάβει διατάξεις, αλλά αυτό είναι το μήνυμα το οποίο και το Συμβούλιο θέλει να ακούσει εν τέλει. Θα δούμε μετά το αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά την ε, ικανοποίηση κοινωνικών κριτηρίων, τι κάναμε, τι δεν κάναμε και είμαστε αντίθετοι στην πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δυσκολεύουμε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Τι κάναμε. Εμείς με δεσμευτικούς νομοθετικούς τρόπους προστατεύουμε το δικαίωμα στην εργασία. Είναι σημαντικό για εμένα. Για τον απλούστο λόγο ότι αυτό που είναι δεσμευτικό, υποχρεωτικό, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο, σαφές, καθιερωμένο, κατανοητό δεν μπορούμε ως υποχρεωτικά κριτήρια να συμπεριλαμβάνουμε αφηρημένες έννοιες. Όταν λοιπόν έχουν οριστεί με συγκεκριμένο τρόπο δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί όπου έχουμε προαιρετικά κριτήρια, κοινωνικά, κοινωνικούς προβληματισμούς, αυτά είναι προαιρετικά που κατ' εμέ ευνοούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντιθέτως από αυτό που λέτε εσείς, ευνοούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τις άλλες, ότι πρώτον εξαλείφουμε το ο κριτήριο της χαμηλότερης δυνατής τιμής, της κατώτατης τιμής και λέμε λοιπόν στις δημόσιες αρχές ότι μπορείτε να λάβετε υπόψη σας και άλλα κριτήρια για να αναθέσετε μια δημοσία σύμβαση και δεύτερον όσοι θα έχουν την ευαισθησία να πούν να, μια μικρομεσαία επιχείρηση καινοτόμο ή μια μικρή επιχείρηση που έχει μια προσέγγιση όσον αφορά τους εργαζόμενου του που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Μπορεί αυτό να λαμβάνεται υπόψη για την ανάθεση μιας δημοσίας σύμβασης. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό για, μόνο για τεράστιες επιχειρήσεις. Μπορούν να εφαρμοστεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πιστεύω ότι αυτό που έχουμε συντάξει, γράψει εδώ, που έχουμε αποφασίσει εδώ στο κείμενο αυτό, είναι ικανοποιητικό. Παρότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που εκκρεμούν, ναι, φυσικά ε, αυτό συμβαίνει σε ε, τόσο μεγάλα κείμενα σε τόσο μεγάλο όγκο εργασίας. Αλλά εν τέλει αυτό που κάναμε ανταποκρίνεται στο στόχο τον οποίο είχαμε ορίσει. Ευνοούμε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι το αντίθετο. Uh, Κύριος Κρόιτσμαν, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοράτσα, Μόλι σα εξήγησαν τι πιστεύουν οι φιλελεύθεροι και η κυρία Γκέμπαρ το είπε, πρέπει να ε, σεβόμαστε τα κείμενα και τους νόμους. Και αυτό πρέπει να ε, το πράττουν και οι μικρές και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Όταν ε, εκχωρείται ένα ελάχιστο μισθό, αυτό πρέπει να τηρείται. Η κυρία Κορατσαμπίλτ λοιπόν ή το είπε. Η διοίκηση πρέπει να αποφασίζει για όλα τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, όπως έχουμε δει, ε, έχουμε διάφορα στοιχεία στα οποία προστίθενται μετά νέα στοιχεία και εν τέλει το όλο πράγμα δεν είναι διαχειρίσιμο. Εμείς ε, θέλαμε να συμπληρώνουμε στοιχεία συνέχεια και ειδικότερα για να διευκολύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει. Θα έπρεπε λοιπόν να πούμε ότι ε, πρέπει να δώσουμε ένα, ένα μήνυμα. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την αμοιβαιότητα για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την αγορά. Αλλά όσον αφορά, ας πούμε, τη Siemens, κατέστρεψε όλη την αγορά, καταστράφηκε όλη η αγορά στην Κίνα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε μια σειρά επιχειρήσεων με παγκόσμια παρουσία που φυσικά ενδιαφέρονται σε αυτό που κάνουμε. Um, Αντίθετα από τον κύριο Κρόιτσμαν, εγώ πιστεύω ότι όλες αυτές οι νομοθετικές πράξεις πρέπει να υιοθετηθούν από διάφορους. Εμείς έχουμε ε, ετοιμάσει και εκθέσεις πρωτοβουλίας και είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία για τους διαγωνισμούς από τις ε, αρχές από μικρούς δήμους και κοινότητες. Η Κομισιόν λέει ότι ένας ευρωπαϊκός διαγωνισμός αυξάνει το κόστος κατά 30.000 ευρώ. Επομένως θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτό το κόστος. Κύριε Έγγελ, είμαι εναντίον της ευθύνης των Δήμων και Κοινοτήτων για το εμπορικό δίκαιο. Αυτό δεν πρέπει να λυθεί στο δίκαιο των αναθέσεων και διαγωνισμών, γιατί έτσι αυξάνεται η γραφειοκρατία για τους Δήμους και τις κοινότητες, τις τοπικές αρχές. Ε, μπορεί επίσης να υπάρξει και ντάμπινγκ στην αγορά μιας άλλης χώρας. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν. Μία κοινότητα, ένα Δήμο πρέπει να μπορεί να αγοράζει ε, υπολογιστέ, αλλά δεν πρέπει να σπάει το κεφάλι του για το πού προέρχονται αυτοί οι υπολογιστέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να προωθήσει την εμπορική πολιτική, αλλά δεν θα πρέπει όμω να είναι υπεύθυνε για μια σειρά από γραφειοκρατικά πράγματα οι δίνικοι κοινότητε. Επίση, μιλήσατε για του υπεργολάβου. Θα ήθελα να διασκεδάσω ένα μύθο που υπάρχει Θεωρούμε ότι στις ε, κατασκευαστικές εταιρείες και στις ε, ε, αναθέσεις εκεί υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι έλεγχοι. Αλλά αυτό δεν είναι λάθος των τοπικών αρχών. Γιατί όποιος ασχολείται, οργανώνει ας πούμε τους διαγωνισμούς, δεν εμπλέκεται άμεσα, δεν κερδίζει, δεν μπορεί να ελέγχει τα πάντα. Ε, δεν μπορούν να πληρώσουν οι δήμοι και οι κοινότητες ε, άμεσα επίσης ε, τους υπεργολάβους. Είναι λάθος αυτή η επιλογή. Υπάρχει αυτό στο κείμενο ως εναλλακτική λύση, αλλά σε αυτήν την περίπτωση εξασθενεί την, τις τοπικές αρχές, οι οποίες πρέπει να σεβαστούν μια σειρά από κριτήρια. Να γιατί δεν συμφωνώ με όλα αυτά. Για τα κοινωνικά κριτήρια έχω διαφορετική θέση από την κυρία Μπίλτ. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι είναι σωστό να πούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη μας τα κοινωνικά κριτήρια. Μπορεί αυτό να, να, μπορεί να ρυθμιστεί μέσω των τεχνικών προδιαγράφων όπως τα περιβαλλοντικά κριτήρια. Θέλω να δώσω τη δυνατότητα στι τοπικέ αρχέ, αλλά όχι να τις υποχρεώσω. Θέλω να του δώσω τη δυνατότητα να εντάξουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στις τεχνικές προδιαγραφές, να προωθήσουν ε, προϊόντα που παράγονται με σωστούς τρόπους, ε, προϊόντα που σέβονται την ευμερία των ζώων, αλλά θα πρέπει να είναι μία επιλογή που έχουν οι τοπικές αρχές, όχι κάτι που τους επιβάλλεται. Επίσης, συμφωνώ σε κάτι μαζί σας ότι υπάρχουν κάποιοι ορισμοί που δεν είναι σαφείς, θα πρέπει αυτοί να ξεκαθαριστούν και θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα κείμενο με ξεκάθαρους ανταγωνισμούς, ώστε να επικυρωθεί, αυτό το κείμενο. Και από τα δικαστήρια. Γιατί αν αυτό το κείμενο μέσω ας πούμε προσφυγών φτάσει στο δικαστήριο θα πρέπει να έχουμε ένα κείμενο με ξεκάθαρους ε, ορισμούς. Ε, δεν θα πρέπει να κινδυνεύουν δηλαδή για λάθος λόγους οι κοινότητες και οι τοπικέ αρχές γενικά να βρεθούν ενώπιον του δικαστηρίου. Έντονη ήταν η συζήτηση. Α, αύριο ψηφίζεται, ούτως ή άλλως δεν θέλω να επιμηκυνώ αυτή τη συζήτηση. Να κάνω ένα-δύο σχόλια. First of all, I think that we're all όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξουν ωφέλη από αυτή την πρόταση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους μικρούς εργολάβους, για τις μικρές αναθέτουσες αρχές, για τις μεγάλες. Είναι μια πρόταση που πρέπει να είναι οπωσδήποτε ευέλικτη, ε, γιατί καλύπτει μια πλειάδα ατόμων και οργανώσεων και φορέων. Θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά, θα πρέπει ε, να, έχουμε, ένα κείμενο ποιοτικό. Ήταν, είναι ποιοτικό το κείμενο, ε, Ευχαριστώ τον Κλάους Βίτε. Τους επόμενους μήνες θα ακούσουμε πολλές παρεμβάσεις από αυτόν στις διαπραγματεύσεις. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στις, στις συζητήσεις μας μέχρι τώρα είναι ότι ενώ έχουμε πολλές τροπολογίες, συχνά ε, καταλήγουμε ότι καμία από τις τροπολογίες αυτές δεν μπορεί να βελτιώσει το κείμενο της Κομισιόν. Ε, και ενώ κάναμε πολλές αλλαγές, η ουσία της πρότασης έμεινε ανέπαφη. Η πρόταση για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και η υποστήριξη καινοτόμων προγραμμάτων, τα νέα εργαλεία για τις ε, ε, εταιρικές σχέσεις ε, για τις προμήθειες είναι προτάσεις που θα χρησιμοποιηθούν πολύ ευρέως από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει αυτό να υπάρχει στον πυρήνα αυτής της πρότασης. Αυτό είναι μία από τις σημαντικές αλλαγές αυτή της πρότασης. Μην το ξεχνάμε ενώ μπαίνουμε σε λεπτομέρειες του κειμένου. Αυτό, αυτό είναι βασικό σημείο για την αμοιβαιότητα. Να σας υπενθυμίσω ότι η νέα πρόταση για την αμοιβαιότητα που υπέβαλε η Κομισιόν, ε, επί της οποίας γνωμοδοτεί ο κ. Σέγγελ ε, και πρόκειται να τα συζητήσουμε ε, στην Επιτροπή, ήδη ενεργοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε τα, τα, ζητήματα της αμοιβαιότητας από την πρόταση αυτή. Η οδηγία για τις 10 είχαν κάποιες ρήτρες για την αμοιβαιότητα. Το να κρατήσουμε αυτά τα θέματα στην βασική οδηγία δεν, α, ούτως ή άλλως δεν ρυθμίζεται οριστικά μέσω της πρότασης για τις ΔΕΚΟ. Επίσης, ε, για την κλασική οδηγία μπορούμε να έχουμε ε, προβλήματα στο Συμβούλιο, αλλά ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά στις διαπραγματεύσεις, σε συνδυασμό με την άλλη οδηγία για τις ΔΕΚΟ. Επομένως, μην τα ξεχνάμε αυτά τα θέματα. Μέσα σε αυτό το πνεύμα ελπίζω όλοι να δουλέψουμε. Και θα δώσω στον κύριο Ταραμπέλα που δούλεψε σκληρά το λόγο για τα τελευταία σχόλια πριν από την αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος μετά τις διάφορες παρατηρήσεις που έγιναν. Και να κρατήσω την ψυχραιμία μου, παρόλο που είναι δύσκολο μερικές φορές και θα σας πω μετά γιατί θα το καταλάβετε. Για την διαδικασία θα τα ξαναπούμε αύριο. Δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Άκουσα τις απόψεις σας, ενδιαφέρον, θα τα πούμε αύριο. Αλλά ας μιλήσουμε επί της ουσίας καλύτερα, για το περιεχόμενο. Η αμοιβαιότητα, αυτά που είπε η κυρία Ρούλη δηλαδή, ποια είναι η συζήτηση, τι διακυβεύεται, είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτεί, τέλο πάντων να προτείνει από τους εταίρους μας να έχει το ίδιο βαθμό ανοίγματο όπως εμείς που έχουμε και θέλουμε να διατηρήσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να αναδιπλωθούμε, θέλουμε να μείνουμε μια ανοιχτή οικονομία. Αλλά συγχρόνω, θέλουμε περισσότερη συνεργασία από τους ε, άλλους φορεί. Να μην έχουν δυσκολίε, οι επιχειρήσει μας δίσδυση στην αγορά. Κοινωνικά κριτήρια. Μην περιπλέκουμε τα πράγματα. Και εδώ, το είπε και ο Έγγελ, υπάρχουν τα υποχρεωτικά κριτήρια, υπάρχει τήρηση των κανόνων, των αρχών και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια κριτήρια που είναι θελοντικά. Μπορούμε εδώ να ενισχύσουμε κάπως την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά μην περιπλέκουμε τα πράγματα. Οι δημόσιες αρχές, όταν είναι δυνατόν, μπορούν να ενσωματώσουν τα κριτήρια. Δεν είναι πάντα εφικτό. Να προσαρμόσουμε το κείμενο, συμφωνώ αλλά μην περιπλέκουμε τα πράγματα. Να δώσουμε στις δημόσιες αρχές την δυνατότητα να κάνουν αυτό που οικονομικά τους συμφέρει περισσότερο με μια ισορροπία. Αλλά να μην τις υποβάλλουμε στη δικτατορία της πιο χαμηλής τιμής. Υπάρχουν τώρα και ευαίσθητα θέματα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Κρότσμα, νομίζω ότι πολύ προσεκτικοί ήμασταν με το πιστοποιητικό για τις δημόσιες συμβάσεις, το ευρωπαϊκό, που δεν θα χρειάζονται πια τόσο βαριές διαδικασίες, τόσα πολλά έγγραφα απριόρι. Θα μπορεί να υποβάλει πρόταση χωρίς τέτοιο βάρος εγγράφων και μετά μπορούμε να απαιτήσουμε τα έγγραφα. Πάμε δηλαδή προς την απλοποίηση. Απλοποίηση επίσης για την κοινή προσέγγιση. Εντάξει, εγώ δεν θα σας αποκαλύψω όλη τη στρατηγική μου, αλλά όταν ε, ξεκινήσαμε από την αρχική πρόταση και φτάσαμε στις μικρές κοινότητες και είπαμε ας τις αφήσουμε να οργανώνονται όπως θέλουν. Ή κάνουν πακέτα ή δεν κάνουν, να το αποφασίσουν εκείνες. Στον Μάρκορν Χάρμπορ τώρα για τη διαδικασία είπαμε, αλλά και ο κύριος Κρόιτσμαν ενδιαφέρεται πολύ για την υπεργολαβία όπως και εσείς, είναι επιθυμητή στις αγορές. Γιατί έτσι επιτρέπει την είσοδο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, όπου σήμερα λίγο συμμετέχουν. Οπότε πρέπει να προτείνουμε στα κράτη-μέλη και αυτό κάνουμε, να μην είναι υποχρεωτικό. Ε, λέμε may, εγώ θα προτιμούσα να λέγαμε shall, θα. Και για να μην το βάλουμε ως δυνατότητα. Αλλά λέμε ότι έχουν τη δυνατότητα δεν θέλουν όλοι να είναι υπεύθυνοι για όλους, αλλά διευκρινίζονται έτσι τα πράγματα. Εντάξει, να τα ξαναδούμε άμα θέλετε, να μπλύνουμε κάπως τις γωνίες, αλλά υπεργολαβία, ε, όταν δεν εφαρμόζεται καλά, αποτελεί ένα παράθυρο για να πετάγονται έξω τα χρήματα και δημιουργείται και κοινωνικό dumping με κατάργηση θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις, στις μικρές κυρίως. Σήμερα στις Βρυξέλλες ε, υπήρχε μια διάδήλωση ε, των ε, εργαζόμενων στον οικοδομικό τομέα και στην ξυλία. Γιατί, γιατί χάνονται θέσεις απασχόλησης, γιατί γίνεται αθέμητος ανταγωνισμός. Και εγώ θέλω να αλλάξει η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, αλλά είναι ένας κανόνας που υπάρχει. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό. Ασχολούμαι με την δουλειά ε, που γίνεται... Ε, κοιτάξτε, στη χώρα μου έχουμε φτάσει να χτίζουμε φυλακές γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Οι Ρωμάνοι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να τηλεφωνάνε στις χώρες τους, οι εργαζόμενοι έτσι, γιατί δεν τους πληρώνανε και έπρεπε να στήσουν λεφτά από τη χώρα τους. Ναι κυρία Ρούλελ, ναι, περιμένετε. Το καλύτερο το αφήνω για το τέλος και είναι το δικό σας. Λοιπόν, τι κάνει η αστυνομία. Θα τελειώσω με την κυρία Ρούλε. Και εδώ είναι που πρέπει να κρατήσω την ψυχραιμία μου γιατί είδα σε τι βαθμό λαϊκισμό, ρήπανση, δεν ξέρω γιατί το κάνετε. Πάντως πριν τις 18 Δεκεμβρίου, πριν την ψηφοφορία τότε, πήρα από το CSRR, το Συμβούλιο δηλαδή ε, Κοινοτήτων της Ευρώπης, τον ανακοινωθέν τύπου, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι εδώ μέσα γιατί δεν ξέρω που βρίσκεται. Εν πάση περιπτώσει, που ε, κατήγγειλε το σχέδιο συμβιβασμού, όχι δεν είναι σεξισμός αυτός, μιλάω για ένα σχόλιο που έγινε πριν την ψηφοφορία και κατήγγειλε το γεγονός ότι βαραίνουμε τη θέση των κινήτων κτλ. Όχι, αυτή είναι διανοητική ρήπανση που έρχεται από την κυρία Ρούλε. Διότι μόλις ανέφερε ψεύδι όταν λέει ότι φορτώνουμε τις κοινότητες. Όχι. Είναι το, κράτος, το κάθε κράτος μέλος από τη δικιά του μέθοδο επιθεώρησης που το κάνει αυτό. Και σαν στις πληρωμές μερικές χώρες τις κάνουν, έχουν κανόνες για να διευκρινίζεται αυτή η αλυσίδα η υπεργολαβής. Μα αφήστε με, εσείς είπατε ανοησίες, αλλά εγώ σας άφησα να τις πείτε. Ε, αφήστε με να μιλήσω κι εγώ τώρα κυρία Ρούλε. Γιατί εσεί παριστάνετε ότι υποστηρίζετε τι μικρέ κοινότητε. Εγώ εδώ και 18 χρόνια είμαι δήμαρχο και έχω ευαισθητοποιήσει. Τη ζωή των κοινοτήτων και το Δήμο τη γνωρίζω πολύ καλά. Και ξέρω ότι είναι ευαισθητοποιημένε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Εμεί θέλουμε να αφήσουμε τι κοινότητε να κάνουν καλύτερε επιλογέ. Το ξέρει και η Επιτροπή και να χρησιμοποιούνται να χρησιμοποιεί το δημόσιο χρήμα πιο αποτελεσματικά. Και μην το λέτε, είναι λάθο να λέτε ότι εμεί θέλουμε να ρίξουμε το βάρο του ελέγχου στι κοινότητε. Όχι, δεν είναι αυτό ο ρόλο του. Υπάρχουν κοινωνικέ υπηρεσίε. Εσεί αναφερθήκατε στην αστυνομία, εντάξει, είναι η ένοπλη δύναμη. Αλλά υπάρχουν κοινωνικέ υπηρεσίε που πρέπει να λειτουργούν καλά. Εμεί ζητάμε από τα κράτη-μέλη να βάλουν πιο ξεκάθαρου κανόνε όσον αφορά τι ευθύνε που έχει ο καθένα, σε αυτή την αλυσίδα υπεργολαβία που ισχύει σε πολλέ χώρε. Όλοι έχουν να κερδίσουν. Δεν είναι επιβαρυντικό για τι κοινότητε αυτό και του δήμου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα για τα οποία δεν θα αναφερθώ, αλλά αυτό, σας λέω αλήθεια, το έζησα πάρα πολύ άσχημα. Τα ακούσατε, μένω ήρεμο, έτσι. Δεν μπορώ όμως παρόλα αυτά να δεχτώ. Δέχομαι την κριτική ευχαρίστω όταν αιτιολογείται, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτά που είπατε και να έρχεται η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ευρώπης και να κάνει τέτοια ανακοινοθέντα σαν και αυτό που έκανε πριν την ψηφοφορία και που δεν ανταποκρίνεται καν στην πραγματικότητα του συμβιβασμού στον οποίο καταλήξαμε. Πρόεδρος. Καλά. Όπως είπα και πριν, ήλπιζα να περάσουμε στην ψηφοφορία αύριο με ήρεμο πνεύμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, εδώ εσείς έχετε διαφορετική άποψη. Ξέρω ότι είναι πολύ ευαίσθητο πολιτικά το θέμα, αλλά υπενθυμίζω ότι πρέπει να έχουμε ηρεμία. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες και αυτό που πρέπει να φροντίσουμε είναι να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να προσφέρει ωφέλη σε όλους. Και πρέπει να ξέρουμε τι θα αποφασίσουμε. Αύριο γιατί βάσει βάση αυτού θα πάμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ελπίζω να μην έχουμε τις ίδιες εντάσεις. Στο Συμβούλιο δεν ξέρω τι θα κάνουν και εκεί οι διάφορα κράτη θα έχουν ε, έντονες απόψεις για το πώς θέλουν να διαχειριστούν τις δημόσιες συμβάσεις για τα αγαθά αυτά. Θα δούμε. Δεχτήκαμε ότι όσον αφορά τη διακυβέρνηση δεν θέλουμε μια βαριά δομή, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε πράγματα στα κράτη-μέλη, θέλουμε μια ελαφρά εντό αγωγικών, light πρόταση. θα πρέπει να αποφασίσουμε όταν συναντηθούμε με τα κράτη-μέλη για το τι ακριβώς θέλουμε. Αφήνοντας ανοιχτή βέβαια την ενιαία αγορά και ενθαρρύνοντας, ενθαρρύνοντας καλές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Έτσι τελείωσε η συνεδρίασή μας. Οι συντονιστές τώρα, παρόλο που βέβαια έχουμε αργήσει. Όσοι δεν θα μείνουν για τους συντονιστές, να εγκαταλείψουν την αίθουσα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και ας προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στη συνεδρίαση των συντονιστών, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας.